Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας ότι πρέπει σιγά σιγά να ξεκινάμε. Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν να υθετήσουμε την μερισία διάταξη, δηλαδή το πρώτο θέμα μας. Υποθέτω ότι δεν έχουμε πρόβλημα και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι 3,5 με 5 θα συζητήσουμε σχετικά με τις ε, θέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 5 με 6 θα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψε με τον νέο πρόεδρο της ομάδος του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον κύριο Τόγερμαν, ο οποίος εκπροσωπεί την EIS και τον καλωσορίζω και από τις 6 έως τις 8 θα συνεχίσουμε ε, διότι γύρισε χθε το βράδυ η αρμόδια επιτροπή από την Τινησία και θα είναι μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμ για να διατυπώσουμε συγκεκριμένες ιδέες για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε την, με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο την επανάσταση στην Τινησία διότι φαίνεται ότι είναι κάτι ανήκουστο, πρωτοφανές και κατά τη γνώμη μου είναι ελπιδοφόρο, επιφέρει όμως και πολλούς κινδύνους. Οπότε δεν ξέρω αν είναι αναγκαίο να το δηλώσω αλλά πρέπει να στηρίξουμε την επανάσταση δεν είναι κάτι που λέμε καθημερινά εδώ τώρα σημείο 2 Υποθέτω ότι μπορούμε ε, να εγκρίνουμε τις, ε, ε, τα πρακτικά της συνεδριάσεως της 30 Σεπτεμβρίου 2010 υιοθετούνται και θα ήθελα εδώ να τονίσω μία τραγωδία η οποία μας πλήττει η περίπτωση του David Κέιτρελ Κισόλε σε μία εβδομάδα όπου έχουμε όλο και περισσότερα ανησυχητικά γεγονότα στον κόσμο πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στην ε, δολοφονία του David ε, Κισόλε ο οποίος ήταν ένας πολύ ενεργός ακτιβιστής και θυμάστε ότι ο Ντέβιτ Κέιτο είχε έρθει επανειλημμένο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, προσφάτως συμμετείχε σε μία κρόαση της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Μικαιωμάτων ε, σχετικά με ε, το AIDS και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πέρυσι ε, το Νοέμβριο αναφέρθηκε εις τον επικίνδυνο ρόλο των LGB στην Ουγγάντα μας έδειξε τις ε, ε, τρομακτικές εικόνες ενός περιοδικού που λέγεται Rolling Stone αλλά δεν είναι το αμερικάνικο το οποίο δημοσιεύει ονόματα και εικόνες για άτομα τα οποία είναι ομοφιλόφιλοι και πρέπει να ε, καταστραφούν και τα κακά νέα της της ε, δολοφονίας του Ντέιβιτ Κέτο μας ε, ε, έφτασαν στις 26 Ιανουαρίου τον σκότωσαν μαζί με τον στο σπίτι του και μαζί με τους άλλους προέδρους των εξωτερικών υποθέσεων και των αρμοδίων επιτροπών ε, διατυπώσαμε ε, ε, τα συλληπιτήριά μας γιατί πολλές φορές είχαμε ανησυχήσει για τους LGBT και στην Ουγκάντα και είχε με ένα ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ελπίζαμε ότι θα μπορέσει να ξαναέρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. LGBT σημαίνει lesbian and gay, bisexual, transsexual people. Λοιπόν, ε, ε, πρέπει να σας πω ότι αφού δείξουμε αυτό το φιλμάκι ε, θα ε, ε, κρατήσουμε ενό λεπτού σιγή για τα, ένα άτομο το οποίο υπεράσπισε τις ιδέες του και θα σας παρακαλούσα να βάλετε τώρα τα ακουστικά σας όλοι για να ακούσετε τι είπε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 Οπότε θα τον θυμόμαστε τον David Κέιτο φαίνεται απίστευτο ότι έχει έρθει εδώ επανειλημμένος και ουσιαστικά είχε έρθει και πρόσφατα και ανησυχούσαμε πάρα πολύ για την ε, επιστροφή του στην ε, πατρίδα του. Ε, Συνεχίζω με διάφορες ανακοινώσεις. Καταρχήν η προσοχή του Γενοβουλίου αυτή την εβδομάδα θα στραφεί προς την Αίγυπτο όπου εντείνονται οι διαδηλώσεις και όπου οι, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναφέρει ότι έχουν σκοτωθεί 300 άτομα, έχουν τραυματιστεί 3.000 και πολλοί έχουν φυλακιστεί. Ε, στην ε, ε, Αίγυπτο σιγά σιγά διακόπτονται όλες οι επικοινωνίες με το εξωτερικό. 30 έως 31 Ιανουαρίου υπήρξαν ε, ε, ε, είσοδοι στις φύλακες και εξήλθαν διάφοροι φυλαξηγισμένοι, ορισμένοι δεν ρώτησαν για τι με αυτόν τον τρόπο έθεσε σε κίνδυνο η κυβέρνηση με την έξοδο των κρατουμένων των φυλακών και ε, εάν δεν μπορούσαν οι πολίτες να χαίρουν ασφαλείας ε, και ε, ηρεμίας. Επιλήφθηκε λοιπόν η Επιτροπή και αποφασίσαμε να στηρίξουμε και τις θεσμικές αλλαγές. Την περασμένη όμως εβδομάδα η Διεθνής Αμνηστία και το, η οργάνωση Human Watch είχε τους ε, εκπροσώπους της οι οποίοι συνελήφθησαν και κρατήθησαν ε, ε, έχω εκφράσει μία, έχω διατυπώσει μία δήλωση καταδικάζοντας αυτές τις κινήσεις ε, ε, γιατί λοιπόν ε, αν στη συνέχεια απελευθερώνονται αλλοδαποί παραμένουν φυλακισμένοι οι Αιγύπτιοι οι οποίοι έχουν παρανόμως κρατηθεί και απαγορεύεται η μετάδοση των ελευθέρων ειδήσεων Πρέπει λοιπόν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα διότι διαφορετικά οι εκπρόσωποι οι οποίοι εμφανίζονται αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να θεωρηθούν σοβαρά εκπροσωπούντες στις δημοκρατικές δυνάμεις. Ε, στη συνέχεια ε, θα έχουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής Μασρέκ και των εξωτερικών υποθέσεων σχετικά με την κατάσταση στην ε, Αιγυπτό και την Τινησία και υποθέτω ότι πολλοί από εσάς θα θελήσουν να συμμετάσχουν. Η τελευταία μου ανακοίνηση αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα διότι ολοκληρώνουμε ε, την ε, πρώτη ε, εξέταση του σημαντικού αυτού χρηματικού μέσου για τα ανθρώπινα δικαιώματα το συρίζουμε και τους προσανατολισμούς τους αλλά διαμέσου των ετών πρέπει να πούμε ότι χρήμα, χρειαζόμαστε περισσότερα the instrument should also focus. και γι' αυτό θα έπρεπε να έχουμε μία συνάντηση με την κυρία Λόχ Μπίλερ και την κυρία Γκάρ. Ε, θα πρέπει δε να ε, εντείνουμε την συμμετοχή μας και γι' αυτό ψηφίσαμε να διατηρήσουμε τη δεύτερη ανάγνωση και να διατηρήσουμε στη δεύτερη αυτή ανάγνωση τις ίδιες τροπολογίες που είχαμε υποβάλει στην πρώτη, ζητώντας να ισχύσει η συνθήκη της Λισαβόνας και να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα εκδημοκρατισμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνω μία νέα ανακοίνωση που αναφέρεται στην επιστολή την οποία λάβαμε από την OMCT, δηλαδή τον Διεθνή Οργανισμό ενάντια, εναντίον των βασανιστήριων και ε, η ε, ελβετική κυβέρνηση εκλήθη να αναλάβει τις ευθύνες της αν W. Bush εμφανιστεί στην Ελβετία όπως προβλέπεται για να προωθήσει το βιβλίο του. Αλλά σήμερα στη συνάντηση που είχαμε τον Γενικό Γραμματέα αυτής της σημαντικής οργάνωσης ελέγχθη ότι η πρόσκληση του W. Bush ε, στην ε, ε, Ελβετία έχει ανακληθεί και ε, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ε, συνθήκες ατιμορρησίας. Δεν ξέρουμε βέβαια ποια θα είναι η συνέχιση αυτού του εγχειρήματο, αλλά πρόκειται για μια σοβαρή οργάνωση η οποία αντιτίθεται στα βασανιστήρια και ε, το θέμα που μας απασχολεί είναι το θέμα των βασανιστήριων. Τώρα ερχόμαστε στο, στην ουσία του θέματός μας σήμερα, δηλαδή έχουμε ένα πακέτο θεμάτων για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η αναθεώρηση ε, αυτού του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ξεκινήσει στη Γενέβη και στον, στη Νέα Υόρκη και λέγεται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο εφέτος. Η Επιτροπή μας ζήτησε μία μελέτη η οποία ε, αναλύει τον ε, ρόλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όταν δημιουργήθηκε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2006 και στη συνέχεια εξετάζει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε αυτή την αναθεωρητική διαδικασία διότι στο παρελθόν ήταν δύσκολο η Επιτροπή αυτή να μπορέσει και το Συμβούλιο να μπορέσουν να υπεραμεινθούν των θέσεών τους στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα όμως που υπάρχει το Συμβούλιο αυτό και ένα ανάλογο διευθυντήριο το οποίο χαιρετίζουμε ε, θεωρούμε ότι ο κύριος Στίν πρέπει να παρακολουθεί εκ του στην κατάσταση. Αλλά επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διότι συμμετέχουν μόνο μεμονωμένα τα κράτη-μέλη, έχουμε και, κριτικά, ε, και ε, άλλα θέματα που πρέπει να μελετήσουμε και γι' αυτό ελπίζουμε ότι σήμερα θα μπορέσουμε να εξετάσουμε τις διάφορες εναλλακτικές μας. Ε, παρακαλώ λοιπόν τον κύριο τη δόκτορα Κάρεν Σμιθ, την δόκτορα, ε, η οποία είναι η υπεύθυνη των ε, διεθνών σχέσεων στο London School of Economics και ε, ε, θα μας παρουσιάσει τη μελέτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επισκόψη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η μελέτη αυτή θα διανεμηθεί στην αίθουσα σήμερα. Η, η ε, κυρία ε, συμμετέχει και ε, σε άλλους οργανισμούς και είναι υπότροφος του ε, Ινστιτούτου Ζωμονέ ναι, εις ε, την στην ε, ε, Ιταλία ε, έχει εξετάξει την πολιτική και έχει συμμετάσχει και δημοσιεύσει και πολλά, πολλές μελέτες. Ε, κυρία Σμίθ, λοιπόν σας παρακαλώ να έρθετε εδώ να μας παρουσιάσετε τα πορίσματα το, της μελέτης σας. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να τις συνοψίσετε σε ένα δεκάλεπτο και στη συνέχεια να έχουμε μία ζωντανή συζήτηση με ε, ε, τα μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Έχω διεξάγει τη μελέτη αυτή σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επισκόψη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το έχω παρακολουθεί στο Συμβούλιο αυτό από όταν καταρτήθηκε το 2006 και έχω εξετάσει την εσωτερική και εξωτερική αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σχετικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι η επιρροή του Συμβουλίου αυτού μέχρι στιγμής ε, είναι ε, Επιτροπή ε, πηρεάζεται καταρχήν από το Ισλαμικό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πιέσει το Ισλαμικό Συμβούλιο να εξετάσει τις μεμονωμένες περιπτώσεις κρατών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα το αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αποδεικνύει ε, ε, το πώς μπορεί να λειτουργήσει ε, σε έναν οργανισμό που είναι τόσο πολιτικοποιημένος και κατακαιρματισμένος αλλά η εξάσκηση επιρροής είναι δύσκολη και επιπλέον έχει ορισμένες αδυναμίες η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η οποία είναι είναι αργή, άκαμπτη και όλα αυτά καταλήγουν εις βάρος της ε, επιρροής Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο εξωτερικό. Τα κράτη-μέλη είναι διαιρεμένα σχετικά με ορισμένα βασικά θέματα και ε, δεν είναι δυνατόν να ε, παρουσιάσει κανείς αξιόπιστα τα δικαιώματα των ατόμων έναντι του Συμβουλίου και επιπλέον ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, μπορέσει καλύτερα να συνάψει συμφωνίες με άλλους οργανισμούς και κράτη γιατί μέχρι στιγμής η δυνατότητα αυτή είναι περιορισμένη. Υπάρχει ένα κενό μεταξύ του τι γίνεται στις Βρυξέλλες και τι γίνεται στη Γενέβη. Δεν είναι είναι συνδυασμένη η πολιτική της αυτή με τις υπόλοιπες εξωτερικές πολιτικές και χρειάζεται να γίνει και μία αναθεώρηση ε, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στους επόμενους μήνες Εκεί διατυπώνονται διάφορες προτάσεις για την ε, ε, λειτουργία του Συμβουλίου και το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν ε, λίγες βελτιώσεις στην κατανομή του φόρτου εργασίας μέσα στα πλαίσια του Συμβουλίου και τα πράγματα είναι πιο προβλέψιμα. Επιτρέπεται να υπάρχει περισσότερος χρόνος για συζητήσεις και αν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει το Συμβούλιο αυτό να επιτύχει περισσότερα αποτελέσματα προτείνω να κάνει το εξής να διακηρύξει σαφώς την αντίθεσή τους εις ε, τις ε, ομάδες οι οποίες στέλνουν πακέτα υποψηφιοτήτων στο Συμβούλιο διότι διαφορετικά ε, δεν είναι δυνατόν να ελέγξει κανείς όταν ένα κράτος συνεργάζεται με το Συμβούλιο στον ελεγκτικό μηχανισμό. Επίσης πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες κατά τρόπον ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν και επιμέρους συζητήσεις κατά τη διάρκεια των γενικών συνελεύσεων θα πρέπει να υπάρχει ένας κώδικας συμπεριφοράς, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα εργαλεία για ε, έλεγχο των καταστάσεων και ε, να υπεραμεινθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση των ε, ψηφισμάτων και των εντολών, να επαναλάβει ότι διακηρύσει την ανεξαρτησία του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τρόπον ώστε να μην γίνει υποχείριο το γραφείο αυτό. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί γενικός ο ρόλος Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιγόντως, διότι οι δραστηριότητες πρέπει να είναι πιο εστιασμένες και ε, να προκαλούν μεγαλύτερη συνένεση για να ενισχυθεί το Συμβούλιο και να μπορεί όντως να προστατεύσει και να προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, θα μπορούσε αυτό να γίνει με ε, καλύτερη πλαισίωση ε, του κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στη Γενέβη. Θα πρέπει επίσης ε, το κλιμάκιο αυτό να είναι καλύτερα ενσωματωμένο στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τρόπον ώστε η ύπατη ε, εκπρόσωπος και ε, η σύμβουλή της να μπορέσουν να στηρίξουν τις θέσεις τους ή στο Συμβούλιο. Οι θέσεις των τρίτων χωρών πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο κατά τους διμερείς διαλόγους μεταξύ ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των στρατηγικών ε, ε, εταίρων της και θα πρέπει να υπεραμεινθεί των θέσεών της στη Γενέβη και να εκφράζει σαν Ευρωπαϊκή Ένωση την ε, ε, ε, την δυσαρέσκειά της εάν δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι αυτοί. Θα πρέπει να συμμετέχει στι συνεδριάσεις συντονισμού, στις συζητήσεις με τρίτες χώρες, κατά τρόπον ώστε να προωθεί κείμενα των θέσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στις διάφορες αντιπροσωπείες. Χωρίς όμως να αντιπροσωπεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διότι αυτό θα μείωνε τον χρόνο ομιλίας στις συνεδριάσεις και θα συνεπέφερε και άλλες άλλες ε, όπως παραδείγματο χάρη σπήρωση των άλλων ομάδων ε, θα μπορούσε λοιπόν ε, να συγκεντρωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο να παρουσιάσει λιγότερες δηλώσεις εν ονόμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και καλύτερα να έχει ένα μήνυμα το οποίο μπορεί να μεταδοθεί από πολλές φωνές δηλαδή από τα διάφορα κράτη-μέλη να προωθεί τις ψηφοφορίες αλλά να σκεφτεί εάν δεν θα ήταν καλύτερο ε, να κατανεμηθούν ε, οι, οι, οι δραστηριότητες αυτές στα κράτη-μέλη. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να είναι και πιο φιλόδοξη και οι στόχοι αυτοί θα μπορούσαν να, οδηγήσουν, να αποτελέσουν έναν εξέχοντα στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν του να παρατηρεί τις ανησυχητικές καταστάσεις θα μπορούσε να είναι πιο δραστηρία και να χρησιμοποιεί διάφορα μέσα για να αντιμετωπίσει τη βία διεθνώς και να μπορεί και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να προωθήσει πιο αποτελεσματικά ε, το θέμα του. Ευχαριστώ κυρία Σμιτ, νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρον που σας ακούσαμε για να δούμε πώς ενδέχεται να ε, ε, παραβλέψουμε τη, και να μην υποφεληθούμε τη δυνατότητα που μας δίνεται να υπάρχει μια ενιαία φωνή στο Συμβούλιο και νομίζω ότι επαναλάβατε πολλές συστάσεις τις οποίες ε, το Κοινοβούλιο έχει ήδη υιοθετήσει στα ετήσια ψηφίσματα και που αναφέρονται στην ανάγκη να εγγυηθούμε την ανεξαρτησία του γραφείου, τις ε, διαδικασίες και ε, επίσης ε, η πρόταση του να είμαστε πιο ενεργοί όσον αφορά τις καταστάσεις των διαφόρων κρατών είναι πολύ χρήσιμη. Εμείς πάντοτε στέλνουμε μία μικρή αντιπροσωπεία στη Γενέβη μεταξύ 16 και 18 Μαρτίου θα πάμε φέτος να συναντηθούμε με όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη-μέλη και τρίτες χώρες εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ειδικού εκπροσώπους και, ως, και ούτω καθεξής για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την κατάσταση. Προτού λοιπόν συνεχίσω θα ήθελα να προτείνω να ακούσουμε την ΕΕΣ. E έχουμε τώρα τον κύριο Τόιερμαν και τον ε, κύριο Γιούς πρέπει να συνεχίσουμε να τους ακούμε και η κυρία Άρβιτσον μήπως θέλει να αναλάβει ε, την, ε, την προεδρία της συνεδριάσεως Εάν συμφωνείτε, καλό τον κύριο Τόιερμαν, ο οποίος μόλις ε, έχει, ε, έχει ε, οριστεί ως πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω ενώπιον σας σήμερα και Πραγματικά χαίρομαι για τη ζήτηση που διεξήχθη το πλαίσιο του Συμβουλίου πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, μόνο μια συνάντηση στο πλαίσιο τη ΚΟΧΟΜ για το θέμα αυτό. Θα σα μιλήσω αργότερα. Η επόμενη θα διεξαχθεί την επόμενη Παρασκευή. Είναι δύσκολο να επικεντρωθούμε μόνο σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αλλά θα σας πω επίσης ποια είναι και τα προγράμματά μας τώρα στη Γενέβη. Έχουμε μπει σε φάση εντατικών διαπραγματεύσεων προτού να περάσει το ζήτημα στη Νέα Υόρκη. Θα ήμουν ευγνώμων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ζήτησε την μελέτη. Θα πρέπει να εξεταστεί αναλυτικά και αυτό σίγουρα θα το συζητήσουμε και με τους συναδέλφους στην Γενέβη και στη Νέα Υόρκη. Ε, συντομία να σχολιάσω μερικά από τα σημεία που αναφέρθηκαν στην παρουσίαση. Μια σειρά από βασικά ευρήματα που και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν πρόκειται για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν εντοπιστεί και, εντοπιστεί και σε διάφορες μελέτες πρόσφατα θεωρούμε ότι έχουν ξεκινήσει μια σειρά από προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι προκλήσεις και να έχουμε μεγαλύτερη επίδοση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Να πω κάτι σχετικά με τις συστάσεις που έγιναν για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Επιδειγμάτων γενικότερα. Τώρα, συμφωνούμε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Γενέβη στο Συμβούλιο Δικαιωμάτων θα πρέπει να απομονωθεί από τα τεχτενόμενα στις Βρυξέλλες είναι κομμάτι του παζλ της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ε, πρέπει να εξεταστεί σε διμερές αλλά και σε πολυμερές επίπεδο. Όταν μιλάμε για την ελευθερία της έκφρασης ε, είναι κάτι το οποίο εξτάζεται και διμερός και πολυμερός. Συμφωνούμε απόλυτα λοιπόν ότι ο συντονισμό πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω και φυσικά το COHOM έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και να διασφαλίσει την ε, σύνδεση με τις βασικές πολιτικές. Ένα από τα εργαλεία που έχουμε είναι να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με περιφερειακές ομάδες εργασίας όταν πρόκειται για περιφερειακά ζητήματα και προβλήματα. Π.χ. η προσέγγιση μας στην Γενέβη σε ό,τι φορά τα δικαιώματα στο Μέση Ανατολή θα το συζητήσουμε όχι μόνο με τους, στο πλαίσιο του αλλά και με συναδέλφους από ε, περιφερειακές επιτροπές. Αυτά που συμβαίνουν στο Συμβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να εξετάζεται συνδυασμό με τα όσα πράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκπροσωπηθεί σε ανώτατο επίπεδο στο Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η κυρία Άστον θα μεταβεί στη Γενέβη στι 28 του μήνα και πριν από μερικέ μέρες ε, μέλη του Συμβουλίου θα έρθουν στι Βρυξέλλες. Επίσης, ε, πρώτη φορά από το 2005 θα υπάρξει ένα Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων με την υιοθέτηση των κάποιων συμπερασμάτων ως εκ τούτου λοιπόν πιστεύουμε ότι θα έχει φτάσει στο ζενήθιο η συζήτηση τόσο σε επίπεδο οικοχώμου όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα πρέπει να βελτιώσουμε τις ε, προσπάθειές μας ε, τόσο σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Συμβούλιο αλλά και στην ε, Βρυξέλλες πρώην ε, επικεφαλής Μισελ Τίλεμανς ε, κατά τη διάρκεια της ε, Βελικής Προεδρίας εξέτασε το ζήτημα και φρόντισε να εντατικοποιήσουμε τις επαφές μας και φροντίσαμε επίσης να θίγουμε πάντα τα ζητήματα των δικαιωμάτων σε διμερές επίπεδο. Οργανώσαμε διάφορες βιντεοδιασκέψεις ε, και άλλες ε, συναντήσεις ε, και τις προσεχείς εβδομάδες, ημέρες θα έχουμε τέτοιες διασκέψεις με, στην Αφρική, με χώρες όπως το Μαρόκο κλπ. Αυτό με οδηγεί επίσης στο εξή. Υπόθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο φασιστική. φυσικά σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ε, αυτό το οποίο απαιτείται είναι να ε, θίγει τα ζητήματα των δικαιωμάτων κάθε φορά που υπάρχει λόγος και ή δυνατόν σε πραγματικό χρόνο. Αλλά πολλά πρέπει να γίνουν προκειμένου να το πετύχουμε αυτό. Επίση η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συμβάλλει και να μπορέσει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιώματα να εξετάζει σε πραγματικό χρόνο αυτά τα ζητήματα. Και με τακτικές και με εκτακτέ συνεδριάσεις ε, και αυτά τα θέματα περιλαμβάνονται φυσικά και στην ε, αναθεώρηση, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα είδος συνασπισμού των ε, δυνητικών υποψηφίων για τις αναχώρα αξιολογήσεις και αυτά καταρχήν είμαστε κατά οποιασδήποτε τέτοια αξιολόγηση, εκτός και αν συνεργάζεται η ενδιαφερόμενη χώρα ούτε μπορούμε να ε, υποβάλουμε κάποιες, ε, να καταθέσουμε κάποιες πρωτοβουλίες ε, με την αρνητική γνώμη της ενδιαφερόμενης χώρας. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι δύσκολο και να έχει παρενέργειες. Θυμάστε την έκτακτη συνεδρίαση για, την, για το Σρι Λάγκα, για παράδειγμα. Και πολύ συχνά έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια ιδέα, υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ των ιδεών της πρώτης του συνασπισμού και της άσκηση δρυμίας κριτικής ορισμένων, κατά ορισμένο χωρό. Θα πρέπει να βρούμε κάποιες ε, ενδιάμεσες λύσεις, κάποια χρυσή τομή στην διαδικασία αυτής της αναθεώρησης. Και δύο ακόμη θέματα σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό και για το πολυμερές έργο, αλλά και για το νέο πλαίσιο θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα μεμονωμένα κράτη την εμπειρογνωμοσύνη που έχουν και να συμμετέχουν πολιτικά στις πρωτοβουλίες μας και να έχουμε στενή συνεργασία μαζί τους. Θα πρέπει και οι μεμονωμένες χώρες να συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των θέσεων και των ε, προτάσεών μας. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει και ενιαία φωνή που θα εκφέρεται μέσω της Προεδρίας, αλλά καλό είναι να προσωπείται η Ευρωπαϊκή Ένωση από όσο το δυνατόν περισσότερες φωνές, δηλαδή από μεμονωμένα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ των δύο, καμία αντίφαση. σα ίσα υπάρχει μια ενισχυμένη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία συνασπισμών και την πρόταση αυτή που ακούστηκε. Πιστεύουμε ότι όχι μόνο για τις συνθήκες της Λισαβόνας, χρειαζόμαστε την ενισχυμένη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γενική Συνέλευση και φυσικά θέλουμε ισχυρό ρόλο και μεμονωμένων χωρών για να στηρίξουν και να ενισχύσουν τα μηνύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναθεώρηση. Ορισμένα από τα σημεία της αναθεώρησης συμφωνούν με αυτά που ακούσαμε προηγουμένως στην παρουσίαση. Εμείς ε, κάνουμε πολλές προσπάθειες και να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αναθεώρηση για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις ε, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να, υπερβούμε τις να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες του. Πριν από δύο χρόνια προσπαθήσαμε και να καταθέσουμε καινοτόμες προτάσεις αλλά και να έχουμε καλύτερο συντονισμό μεταξύ μας. Και πολλές χώρες μέλη ξεκίνησαν διασυνοριακές ομάδες και δεσμεύσεις και πρότειναν καινοτόμε ιδέες για τη βελτίωση της θέσης ορισμένων χωρών, για την θέσπιση κάποιων δικτών ενεργοποίησης κτλ. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, ικανότητα του Συμβουλίου να αντιμετωπίσει οι ιδιαίτερες καταστάσεις, το θέμα των διαδικασιών, το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, υπάρχει κάποια ισχυρή αντίσταση αυτή τη στιγμή για την ενίσχυση όλων αυτών των στοιχείων στο έργο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αντιμετωπίζουμε στη Γενέβη με αρκετά δυσχερή διαπραγματευτική διαδικασία. Σήμερα μόλις μας έστειλαν τη, τα πρώτα πρακτικά από, την, από τις διαπραγματεύσεις ε, στη Γενέβη για την, ανα, για την αναθεώρηση και σήμερα παρουσιάσαμε τα εκτεταμένα σχόλια σε ό,τι αφορά την συμπίληση, αυτή πρώτη συμπίληση των συζητήσεων εκεί στη Γενέβη και σε ό,τι αφορά και τις ε, αντιπροσωπείες και τον πρόεδρο θα πρέπει η διαδικασία της Γενέβης να μην περιορίζεται μόνο στις μεθόδους ή στο πρόγραμμα εργασιών του Human Rights Council, αλλά και σε άλλες πτυχές που αφορά τις καταστάσεις των χωρών. Η διαδικασία της Γενέβης είναι το πρώτο βήμα. Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις στη Νέα Υόρκη που θα περιλάβουν και θέματα όπως την ποιότητα της ε, ιδιότητας του μέλους, αλλά και άλλες, ε, άλλες παρατηρήσεις που αφορούν την κατάσταση των χωρών. Σας ευχαριστούμε κύριε Τόιμαν. Κύριε Χέρτς, μήπως θέλετε να συμπληρώσετε την γνώμη του οργάνου που εκπροσωπείτε. Όχι, ανήκουμε στην ίδια ομάδα, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Χαίρομαι που είσαστε μέλος της, αυτής ομάδας και τώρα είναι Άρβινσον, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πολλές, ε, μάλλον οι περισσότερες καλές ιδέες παρουσιάστηκαν από την κυρία Σμιθ στην ομιλία της που ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουση. Θα αναφερθώ σε μερικές ε, από τις βασικές ιδέες ε, της αναθεώρησης. Έχουμε κυκλοφορήσει το έγγραφο το οποίο έχουμε ετοιμάσει και εμείς αλλά και η ειδική υπηρεσία. Τώρα δύο σύντομα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα είπε και, ο, και η κυρία Σμίθ ότι επιθυμούμε τα Συμβούλια των Δικαιωμάτων να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις έκτακτες καταστάσεις ε, και σε, να αντιδράσει σε άμεσο χρόνο, σε πραγματικό χρόνο. Θα ήταν καλό να χρησιμοποιούν ε, τα πάνελ όχι μόνο κατά των συνόδων αλλά και στην περίοδο ανάμεσα στην διεξαγωγή των συνόδων. Και να υπάρχει και μια διάδραση με, ε, με την περιφέρεια. Παρουσιάστηκε η ιδέα ότι το Συμβούλιο μπορεί να οργανώνει έκτακτες ε, συναντήσεις χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα από τις δράσεις που έχει αναλάβει. Δεύτερον, στις ειδικές διαδικασίες ε, η ανεξαρτησία είναι ένα θέμα κλειδί για μας και τρία σημεία σχετικά. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι φορά τον κώδικα συμπεριφοράς, θεωρούμε ότι η εφαρμογή παρόμοιου κώδικα θα πρέπει να οριστεί από αυτορυθμιζόμενα σώματα, ομάδες, να υπάρχουν δηλαδή μελέτες ομοτήμων δεύτερων. Θεωρούμε ότι καλό θα ήταν να υπάρχει και μια αντικειμενική αξιολόγηση των κρατών σε ό,τι φορά την συνεργασία τους θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε λοιπόν αν θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια αξιολόγηση από ένα μηχανισμό και ένα τεχνικό ζήτημα. Το τρίτο, κατά διάρκεια των συνόδων λόγω έλλειψης χρόνου, οι ειδικέ διαδικασίες έχουν προβλεφθεί και η δυνατότητα διάδρασης με τα μέλη είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν ε, ωφελεί στην όλη συζήτηση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια συζήτηση που θα αφορά τον εισηγητή και τους εμπειρογνώμονες πάνω στο θέμα αυτό. Τέλος, για τη δική μας ανεξαρτησία να τονίσω ότι για μας είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Χρειάζεται η Κομισιόν να ενημερώνει το Συμβούλιο για τις δράσεις της. Αν χρειαστεί μπορώ να μπω και σε λεπτομέρειες. ευχαριστώ πολύ κύριε Άρβινσον. Και τώρα ο λόγος στους ε, συναδέλφους, ε, η κυρία Λόχ Μπίλερ, που είναι μέλος, του, μέλος της ομάδας των Εθνών και έχει συμμετάσχει σε πολλές εργασίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον κύριο Σμίθ για τη μελέτη του. Σίγουρα θα πρέπει να την, ε, την κυρία Σμίθ μάλλον, θα πρέπει να την μελετήσουμε διεξοδικά για να την αντιληφθούμε σε όλες τις διαστάσεις. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντα συγκεκριμένες εντολές και ψηφίσματα για χώρες, ακόμη και αν αυτό είναι το πιο δύσκολο. Γιατί δεν ξέρω τι άλλο από τη δομή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μπορεί να φέρει πραγματικά τους παραβάτες ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώπιον των ευθυνών τους. Μόνο αν μιλήσουμε για κάθε χώρα συγκεκριμένα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει είπαμε, να θυγραμιστεί με το έργο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Μέχρι στιγμής είχαμε μία μόνο τέτοια σχετική εμπειρία. Με τη σύνταξη της γνωμοδότησης για τη Frontex, για, την, για τον οργανισμό δηλαδή των συνόρων. Και εκεί είναι εύκολο να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οργανισμοί της θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την τεχνογνωσία, αλλά και το κύρος θα έλεγα, της εμπειρογνωμοσύνης του γραφείου του είπα το αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και όταν προβαίνει σε κρίση για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιτόπου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γραφείο του υπαταρμοστή. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Αναφέρεται το γραφείο του Υπατοαρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν αναφέρονται ε, άλλα τέτοια όργανα. Ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο καλό θα ήταν να υπογραμμίσουν ότι αυτή η τεχνογνωσία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Δεν χρειάζεται να επικαλύπτουμε τις δομές που υπάρχουν ήδη στα Ηνωμένα Έθνη. Επίσης, είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως μπλοκ. Ίσως θα πρέπει να μην επικεντρώνει τις προσπάθειές της στο να προσπαθεί να συσπυρώσει τα κράτη-μέλη. Αυτό για πρώτη φορά το ακούω. Γιατί εμείς ε, στη Γενική Συνέλευση διαπίστωσα ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση χάσαμε ένα ψήφισμα που διεκδικούσε τα περισσότερα ενισχυμένα δικαιώματά μας για να εκπροσωπούμαστε και να εκφέρουμε ενιαία στάση και φωνή. Αυτό συνοδεύει μία ισχυρή και ενεργό διμερή δράση. Αυτά τα διέκρινα από την παρουσίασή σας και όχι από την έκθεση γιατί δεν διάβασα ακόμη, αλλά έρχεται σε αντίφαση με τη δική μας προοπτική που είναι υπέρ της συνένωσης ε, και της συσπήρωση των κρατών μελών για να αποφέρονται με νέα φωνή. Τα μπλοκ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι πολύ ισχυρά και ως ανασχετικές ε, δυνάμεις. Αλλά η Αίγυπτος ήταν πολύ ισχυρός παράγοντας και οι κυβερνήσεις πέφτουν, οι διπλωμάτε μένουν. Και ελπίζω βέβαια στην Αίγυπτο να μην παραμείνουν μόνο ε, οι διπλωμάτες και να αλλάξουν οι πολιτικές, αλλά να αλλάξουν ε, και οι στάσεις ε, ορισμένων χωρών όπω της Αιγύπτου για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζω έτσι να μην αποδυναμωθεί θέση κάποιων ομάδων που είναι κατά των ειδικών ψηφισμάτων κατά μεμονωμένων χωρών. Προς το παρόν δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Ας ακούσουμε την ε, δόκτωρα Σμίθ να θέλει να σχολιάσει, να απαντήσει. Ευχαριστώ. Um, δεν θα πρότεινα να εξαφανιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά ο ρόλος που διαδραματίζει σε ό,τι αφορά να ε, αντιδρά ακόμα και σε κάποιες δηλώσεις ε, κρατών του Νότου, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ε, ωφελεί. Είναι δύσκολο λοιπόν να μπορέσουν κάποιες χώρες να ξεφύγουν από το μπλοκ στο οποίο ανήκουν από τον ε, συνασπισμό ειδικά σε ό,τι αφορά τα ψηφίσματα και τον τρόπο ψήφισης. Λοιπόν, ε, περίπτωση λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μειοψηφία όπως συνέβη με την ε, Σρι Λάγκα. Η ΤΑΤΕ Είναι δύσκολο λοιπόν ε, να κερδίζει κάποιες ψηφοφορίες διότι βρίσκεται σε μειοψηφία. Όπως σας είπα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη. Λοιπόν, Τώρα, για το πώς η Ευρώπη μπορεί να δραματίσει σημαντικότερο ρόλο, αλλά και το πώς τα κράτη-μέλη μπορούν να οδηγήσουν σε μια καλύτερη διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Δικαιωμάτων και να καταστήσει το Συμβούλιο αυτό πιο αποτελεσματικό, θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση των μπλοκ. Είναι αδύνατον η Ευρώπη να δημιουργήσει συνασπισμούς με άλλα μπλοκ στις περισσότερες περιπτώσεις. Εάν τα μπλοκ παραμείνουν όσο έχουν, τότε είναι δύσκολο να <clears throat> υπάρξει βελτίωση των εργασιών του Συμβουλίου. Θα ήθελα να συστήσω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να συντονιστεί αποτελεσματικότερο να θέσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ως μία από τις προτεραιότητες και έτσι πίσω από τις ε, ή και πριν από την διεξαγωγή των συνεδριάζων θα πρέπει λοιπόν αυτός ο συντανισμός να είναι πολύ πιο ισχυρός και αποτελεσματικός. Χρειάζεται λοιπόν τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να οργανωθούν αποτελεσματικότερα και έτσι μερικές φορές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Πολλές φορές οι Ευρωπαίοι είναι αυτοί που οδηγούν τις συζητήσεις, αλλά Εάν δεν μπορέσουν να προωθήσουν αυτή την ενισχυμένη συνεργασία, τότε τα αποτελέσματα θα είναι τα γνωστά. Χρειάζεται λοιπόν να δώσουμε, να βάλουμε μάλλον τις προτεραιότητες. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνήθως ε, λαμβάνουν πρώτοι το λόγο. Αλλά όπως είπα, είπα και προηγούμενα και επαναλαμβάνω ότι αυτή η κατάσταση με τα μπλοκ, με τους συνασπισμούς δεν οδηγεί πουθενά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να οργανωθεί καλύτερα, να συντονιστεί καλύτερα, αλλά και να παρουσιάζει τα ζητήματα με τρόπο ουσιαστικότερο και αποτελεσματικότερο. Αυτά νομίζω θα μπορούσαν να βοηθήσουν το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστούμε, Δόκτωρα Σμιθ. Αυτό που μου έρθει στο μυαλό είναι η ερώτηση μήπως θα μπορούσατε να διευκρινίσετε την ανάγκη της ε, ενσωμάτωσης της θέσης ε, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα ή και οι συνάδελφοι που μίλησαν έχουν υπόψη κάτι τέτοιο γιατί αλλιώς δεν είμαστε ούτε έξυπνοι ούτε αξιόπιστοι αν δεν γνωρίζει αριστερά τι πει δεξιά. Και δεν ξέρω ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτό το θέμα το, της εξωτερικής δράσης. Αυτό που αποκαλούμε στην αναπτυξιακή συνεργασία είναι η ο συνδυασμός των πολιτικών. Και εμείς ε, δώσαμε μάχη για να έχουμε μια τέτοια ενσωμάτωση και λήψη υπόψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι καθόλου εύκολο. Βέβαια διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση και κάτι που παλιά ήταν όνειρο τώρα αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά. Μήπως λοιπόν θα μπορούσατε να απαντήσετε αλλά Πρώτα θα ακούσουμε τον κύριο Πρόντι και μετά τους συναδέλφους από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σύντομα. Δύσκολα μπορώ να κατανοήσω την θέση της κύρια Σμιτ διότι αν ε, δούμε την κατάσταση στην Αφρικανική Ένωση είναι οι διαφορετικές θέσεις των κρατών μελών που καθιστούν δύσκολη την συμφωνία ενώ θα ήταν προς το συμφέρον όλων και για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Αφρικανική Ένωση να μπορεί να ανταποκρίνεται και να απαντά αυτονόμως επί των ζητημάτων αυτών. Δεν βλέπω λοιπόν καμία αντίφαση. Θεωρώ ότι αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να προχωρούν χέρι-χέρι. Μία φωνή λοιπόν για να μπορούν να δημιουργούνται και συμμαχίες και που θα λαμβάνει υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα. Θεωρώ λοιπόν ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να διαδραματίσει ύψιστο ρόλο σε αυτή την δράση σύγκλησης και θεωρώ ότι αν κατορθώσουμε να φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση, τόσο το καλύτερο για όλους. Πρώτα απ' όλα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά θα ωφεληθούν. Εγώ θα έλεγα πως δεν θα πρέπει να το θεωρήσουμε ως αντίφαση, αλλά τον αντίον να φροντίσουμε να ενδυναμώσουμε όλες τις δυνάμεις που συμμετέχουν προς την αυτή κατεύθυνση, διότι μπορούμε να δημιουργήσουμε έτσι μια συνέργεια πολύ σημαντική. Ευχαριστούμε κύριε Πρόντι. Χρειαζόμαστε πιο διεξοδική ανάλυση αυτού του παραδόξου, τουλάχιστον φαινομενικά παραδόξου. Ο κύριος Τόιρμαν. Όντως, πολύ συχνά συναντούμε τέτοιο προβληματισμό. Δεν λέω να εγκαταλείψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη των Ηνωμένων Εθνών. Βέβαια, η συνθήκη τη Λισαβόνα δεν ισχύει στη Γενέβη, στη Νέα Υόρκη, σε άλλη πολυμερή φόρα. Θα πρέπει να βελτιώσουμε όμω πρώτα εσωτερικά τις επιδόσεις μας στη Γενέβη, να, να πραγματοποιήσουμε πιο αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ μας, ενώψε διαπραγματεύσεων στη Γενέβη και αυτό θα πρέπει να το επεξεργαστούμε πρώτα μεταξύ μας και για τα πολιτικά θέματα θέλουμε ενεργό και ισχυρό ρόλο και των μεμονωμένων χωρών. Γιατί ξέρετε πώς ισχύει ο καταμερισμός των ευθυνών στα Ηνωμένα Έθνη και αλλού. Θέλουμε αυτό το θέμα να το προβάλλουμε, να ενισχύσουμε τον, την ενεργό συμμετοχή και μεμονωμένων χαρών μέλων. Και συλλογικά να βελτιώσουμε το συντονισμό μας, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε καινοτόμε προσεγγίσεις. Μία τέτοια καινοτόμα προσέγγιση είναι ένα μήνυμα, αλλά πολλές φωνές. Και αυτό στο πλαίσιο τη αναθεώρηση ε, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαπιστώνουμε ότι ήταν καλέ οι επιδόσει Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δείτε το συνοπτικό έγγραφο, βλέπετε πόσες, πόσο λίγε είναι οι προτάσει μα που ε, λαμβάνονται υπόψη. Επίσης βλέπουμε διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας. Πρόσφατα είχαμε μεγάλη επιτυχία σε διαφορά της Ευρωπαϊκής ευρωπαϊκές για την θανατική ποινή στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά το, τις διασυνοριακές συμμαχίες, και εκεί είχαμε επιτυχία. Αλλά και για τα θεματικά ζητήματα, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, διαφιλικών, αφωτεροφιλοφίλων κτλ. Εκεί επίσης ε, πρωτοστατήσαμε στην ανάληψη πρωτοβουλειών και ε, υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες. Θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω το σύστημα και οι διασυνοριακές συμμαχίες είναι πιο δύσκολες όταν έχουμε μεμονωμένες ε, χώρες, κατάσταση για, μεμονω, για συγκεκριμένες χώρες. Εκεί είναι δύσκολο να εντοπίσουμε, να εντοπίσουμε χώρες στην Αφρική ή την Ασία όταν θέλουμε να ασχοληθούμε με τη ειδική κατάσταση που επικρατεί σε συγκεκριμένες ζώνες της Αφρικής ή της Σε ό,τι αφορά την ατμόσφαιρα που ισχύει στη Γενέβη στο, στα Συμβούλια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από ότι στη Γενική Συνέλευση που εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Μερικές φορές είναι πιο εύκολο να προβάλλουμε κάποιες καταστάσεις ή πρωτοβουλίες στο ένα φόρουμ πιο έντονα από ό,τι στο άλλο, στη Γενική Συνέλευση από ό,τι στη Γενέβη, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και ως προς το τελευταίο σας σχόλιο, η κυρία Λόχμπίλερ είπε τι γίνεται σε περίπτωση μεταστροφής μιας χώρας ε, στη στάση της, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γιατί τη μια μέρα η Αίγυπτος, για παράδειγμα, μπορεί να είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Συμβούλιο και μετά να αλλάξει γνώμη. Εμεί θέλουμε να ενισχύσουμε τη δυνατότητα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να αντιμετωπίσει την κατάσταση συγκεκριμένων χωρών. Και μάλιστα κάποιες χώρες στο Νότο που ήταν ε, υπέρμαχοι ε, στην περιοχή τους, στη ζώνη τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ε, απρόθυμες να το θέσουν πιο σφαιρικά το ζήτημα αυτό στα Ηνωμένα Έθνη. Εμείς προσπαθούμε σε συνεργασία με τους στρατικούς μας εταίρους να φέρουμε στο επίκεντρο το, του πλαισίου και των Ηνωμένων Εθνών τα ανθρώπινα δικαιώματα. Uh, ε, θα ήθελα να απαντήσω την ερώτηση την οποία κάνατε σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ε, ένταξή του σε ένα σύνολο. Δεν πρόκειται απλώς ε, για ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και για το πόση προτεραιότητα δίνουμε στο θέμα αυτό και ενδεχομένως δεν θέλω να υπησέλθω σε λεπτομέρειες αλλά θέλουμε να δούμε ε, ποιες είναι οι άλλες προτεραιότητες μας δημοσίων σχέσεων στην οποία περίπτωση Νομίζω ότι αν κοιτάξετε ποιος στηρίζει τους Ευρωπαίους στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ποιος ψηφίζει με το μέρος τους και ποιος όχι, θα τρομάξετε. Υπάρχουν ε, πάρα πολλές δημοκρατίες και ακόμη και αν γίνει δημοκρατική η ε, Αιγυπτός δεν είναι προφανές ότι θα ε, κλείνει προς την Ευρώπη. ενδέχεται να υπάρξουν ή προς τον δυτικό κόσμο. Υπάρχουν πολλές ε, δίθεν δημοκρατίες ε, ε, σε πολλά σημεία του κόσμου νοτίως και ανατολικά. Οπότε πρέπει να γίνει μία ορθολογιστική συζήτηση για την κατάσταση των χωρών μέσα στα συμφραζόμενά τους απαντώντας σε πολλά ερωτήματα κατά τρόπον ώστε ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιστήσει στην προσοχή των ομολόγων της ότι παρακολουθεί το τι γίνεται στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διότι διαφορετικά ε, ε, ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες έχουν συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνουν ε, γενναιόδερα χέγγια και από την άλλη μεριά την κατακρίνουν στο Συμβούλιο του Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δεν παίρνουν το μέρος της. Εάν λοιπόν ε, δεν υπάρξει ένας διάλογος ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και ε, των στρατηγικών ομολόγων της τότε θα δούμε ότι οι θέσεις αυτές είναι σημαντικές δεν είναι κάτι το οποίο είναι μία φιλική κίνηση ε, δηλαδή να μην υπερψηφίσει κανείς ε, ένα ψήφισμα για τη Σρι Λάνκα όπως έγινε σε μια συνεδρίαση ε, ή ε, ε, ε, θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα διότι τα ψηφίσματα μη δράσεως στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως στην Κίνα σημαίνει ότι σταματάει η συζήτηση επί ενός θέματος και βλέπουμε ότι στηρίζονται από χώρες οι οποίες είναι αρκετά στενά συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν η θέση αυτή να ενσωματωθεί σε ένα σύνολο. Θα πρέπει στη Γενέβη να γίνει μια συζήτηση και να δούμε ε, αυτά τα οποία συζητώνται εδώ στις Βρυξέλλες με τις τρίτες ε, χώρες πώς εντάσσονται σε ένα σύνολο στη Γενέβη διότι πιστεύω ότι όλα αυτά είναι σημαντικά στοιχεία της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι σύντομα θα τελειώσει αυτή η συζήτηση και δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Λοχμπίλερ. Ευχαριστώ. Ε, θα είναι πολύ σύντομη η παρατήρησή μου, αλλά και είπατε κυρία Σμιθ ότι υπάρχουν στενοί δεσμοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμήθηκα λοιπόν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και όλες τις γραμμές επικοινωνίας με το Κογκρέσο στις Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων ήταν σαφέστατη. Δεν θυμάμαι σε ποιο περιοδικό σημαντικό και είπε ότι αν το Συμβούλιο Ανθρωπίνων ε, Δικαιωμάτων ε, δεν ε, προσφέρει αυτά τα οποία θα έπρεπε τότε γιατί θα το χρηματοδοτεί οι Ηνωμένε Πολιτείε. Οπότε αν συσπηρωθούμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρχει μια πιο ενεργή συμμετοχή και αν δεν παραμείνουμε όπως το παρελθόν παρατηρητές. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γυρίσουμε σελίδα. Βέβαια παραμένουμε σε αρμοδιότητες ε, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Αθηνών και περάμε στο σημείο 5 που έχουμε τη συνέχεια της έκθεσης Stone σχετικά με τις συγκρούσεις της Γάζας και την έκθεση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Αθήνων σχετικά με το επεισόδιο με το στολίσκο που έπλε προς τη Γάζα. Όπως συμφώνησαν οι συντονιστές της υποεπιτροπής μας, προσπαθήσαμε να προσκαλέσουμε τον ίδιο το δικαστή Goldstone στη συνεδρίασή μας, αλλά δυστυχώς ε, ακολύεται. Παρακαλώ, οι ιδιωτικές συνομιλίες ε, να γίνονται εκτός αιθούσης. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο δικαστής Goldstone μας ανακοίνωσε μέσω του γραφείου του ότι πολύ ευχαρίστως θα συμμετείχε σε ανταλλαγή απόψεων στο μέλλον, σε κάποια συνεδρίαση που θα βόλευε και τον ίδιον, Αλλά έχουμε δύο εκπροσώπους ε, της ε, Επιτροπής που επίσης δεν μπόρεσαν να έρθουν σήμερα για εξαιτία ανηλυμένων υποχρεώσεων τους, αλλά έχουμε τον κύριο Άρβιτσον, την κυρία συγγνώμη Άρβιτσον, που θα μας ενημερώσει ως προς τις τελευταίες εξελίξεις Έχετε λάβει σχετική τεκμηρίωση, αγαπητοί συνάδελφοι, και στο χαρτοφυλάκιο σα αλλά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λάβατε και την ίδια την έκθεση Goldstone. Θα έδωσω το λόγο 8 λεπτά στον κάθε προσκεκλημένο. Πρώτα στην κυρία Άρβιτσον, κατόπιν στον Τάρεκ Μάρι, από το Διεθνές ε, Νομικό Γραφείο της Παλαιστίνης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην κυρία Μίρι Βαν Κάρτεν, την τρίτη προσκεκλημένο μας που είναι ε, ακτιβίστρια Ισραηλινή και μάλιστα συμμετείχε σε μία οργάνωση ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ισραήλ. Καλώς ήρθατε και οι τρεις. Οκτώ λεπτά ο καθένας παρακαλώ. Πρώτα η Λίνα Άρβιτσον. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία στις τελευταίες εξελίξεις, τι συνέβη μετά την υποβολή των διεκθέσεων, την έκθεση της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής του ΙΕ για τα επεισόδια στη Γάζα, την έκθεση Goldstone, αλλά και την ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ που διερεύνησε τις σοβαρές παραβιάσεις ε, σε ό,τι αφορά την απομπή που έπλεε στη Γάζα, τη γνωστή έκθεση για το στολίσκο δηλαδή. Έκθεση Goldstone υπευλήθη το Σεπτέμβριο του 2009 στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στις 574 σελίδες της η έκθεση Κολστόν περιέλαμβανε ανάλυση 36 συγκεκριμένων επεισοδίων στη διάρκεια συγκρούσεων της Γάζας στην περίοδο 2008-2009 και κατέληγε στο συμπέρασμα ότι και Ισραηλές και Παλαιστινιακές Ένωπες Δυνάμεις ε, διέπραξαν ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και ενδεχομένως και εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης στη Γάζα και ζήτησε και από τις δύο πλευρές να διενεργήσουν αξιόπιστες και αντικειμενικές έρευνες. Η ΔΕΜΗ θα έπρεπε τα ζητήματα αυτά και οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και εγκλημάτων πολέμου να παραπευθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Τι συνέβη έκτοτε. Το 2010 το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγκρότησε μια νέα ανεξάρτητη επιτροπή που ανέλαβε την αποστολή της παρακολούθησης και αξιολόγηση οποιασδήποτε χώριας δικαστική ή άλλης διαδικασίας του Ισραήλ ή της Παλαιστίνης για τη διερεύνηση των επεισοδίων που επεσήμανε η έκθεση Goldstone. Η Επιτροπή αυτή παρακολούθησης υπέβαλε την πρώτη της έκθεση πριν από λίγους μήνες, στην οποία κατέληγε στα εξή συμπεράσματα. Καταρχήν, το Ισραήλ διενήργησε κάποιες ε, έρευνες για πολλά επεισόδια, μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις όμως ε, απήγγειλε κατηγορίες και μάλιστα σε μία περίπτωση είχαμε και καταδίκη για κλοπή πιστοτικής κάρτας. Δεύτερον, οι έρευνες δεν, κατέλ, δεν περιλάμβαναν όλες, όλα τα επεισόδια που επεσήμανε η έκθεση Goldstone. Επίσης, ε, το Ισραήλ δεν ε, επέκτηνε τις έρευνες σε υψηλούς αξιωματούχους, ούτε ερεύνησε ισχυρισμούς για παραβιάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Όχθη ε, που επεσήμανε η έκθεση ότι είχαν διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης. Επίσης, ε, εκφράστηκαν ανησυχίες για το κατά πόσο όντως ήταν αμερόληπτη η διεξαγωγή της έρευνας από Ισραηλινής πλευράς. Η Επιτροπή αυτή παρακολούθησε και αξιολόγησε και τι έρευνε που έγιναν από Παλαιστινιακής πλευράς σε ό,τι αφορά τις έρευνες ε, της Παλαιστινιακής Αρχής, η Επιτροπή αυτή παρακολούθησης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Παλαιστινιακές Αρχές ε, συγκρότησαν ανεξάρτητη ερευνητική επιτροπή και μάλιστα συναντήθηκε με τα μέλη της Επιτροπής αυτής και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ε, οι έρευνες που διεξήχθησαν από την Παλαιστίνη πληρούσαν τις διεθνείς προδιαγραφές. Βέβαια, δεν ε, διερευνήθηκαν πλήρω οι ισχυρισμοί για σοβαρές παραβιάσεις ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, δικαιωμάτων, ε, και εγκλημάτων πολέμου στην ζώνη της Γάζας εξαιτία προβλημάτων πρόσβασης στην Γάζα. Η Διερευνητική Επιτροπή που συγκροτήθηκε από τη Χαμάς συνάντησε μέλη και τον και της Επιτροπής ε, ε, της Ad Hoc Επιτροπής Παρακολούθησης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν διερευνήθηκαν επαρκώς οι ισχυρισμοί της έκθεσης Goldstone. Στο μεταξύ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανανέωσε την εντολή αυτή τη Επιτροπή Παρακολούθηση και μάλιστα μόλι πρόσφατα συνέχισε το έργο τη με δύο ανεξάρτητου εμπειρογνωμόνε, τη δικαστή Μακαβεν Ντέβι και την δικαστή ε, Άσπερ Μαγκάουν. Στόχος ήταν να αξιολογηθούν οι πρόσφατες έρευνες που έγιναν από τις δύο αρχές και επίσης ε, να πραγματοποιηθεί μια αποστολή στην περιοχή προκειμένου να γίνουν συνομιλίες με ενδιαφερόμενους ε, και αρμοδίους για ενημέρωση ως προς την ε, περιοχή. Μάλιστα, κατά πάσα πιθανότητα η ενημέρωση θα γίνει στις 21 Μαρτίου στη συνέλευση και τότε θα γνωρίζουμε και τα πορίσματα αυτής της ε, Επιτροπής. Σε ό,τι φορά την έκθεση για το στολίσκο, η έκθεση για το στολίσκο της Γάζας ε, καταρτίστηκε από μια τριμελή διερευνητική αποστολή που συγκροτήθηκε δύο μέρες μετά το επεισόδιο, στις 2 Ιουνίου του 2010. Ε, δικαστής Κορλ Φιλίπς από το Σερντές Σίλβα πρώην εισαγγελέα της, ε, του Ειδικού Δικαστηρίου της Ιεραλεόνε και Μέρια Τάρια πρώην μέλος της Επιτροπής για την κατάργηση διακριτικής μεταχείρισης βάρος των γυναικών. Αυτή η, η Επιτροπή ε, έκανε με 112 μάρτυρες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παραβάζει διεθνούς δικαίου καθώς και διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαπράχθησαν από το Ισραήλ και στα πλοία του στο Λίσκο, αλλά και κατά τη διάρκεια της κράτησης ε, των μελών της ε, νεοπομπής στο Ισραήλ. Επίσης, ε, περιλαμβάνονταν στην έκθεση αυτή και κάποια πορίσματα σε ό,τι αφορά την, μεταχείριση ή τη συμπεριφορά μάλλον στρατιωτικών και μάλιστα έξι από τους εννέα θανάτους οφειλόταν σε συνοπτικές εκτελέσεις. Επίσης διαπιστώθηκε μία απαράδεκτη συνέχιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα εξαιτία ε, συλλογικών τιμωριών. Η έκθεση αυτή περιλάμβανε κάποια ανάλυση πραγματικών παριστατικών, αλλά δεν περιλάμβανε και συστάσεις. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέτασε την έκθεση πριν από δύο μήνες και ε, ζήτησε από τον ύπατο αρμοστή να ζητήσει συνέχιση αυτής της έκθεσης ε, στην επόμενη συνέλευση του Μαρτίου. Μάλιστα, η Επιτροπή αυτή ζήτησε πληροφορίες από το Ισραήλ, την Τουρκία και την Παλαιστινιακή Αρχή για τα βήματα που πραγματοποίησαν οι αντίστοιχε κυβερνήσει για να δώσουν μια συνέχιση σε αυτή, σε αυτή την έκθεση και μάλιστα η σχετική ενημέρωση θα γίνει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Μάρτιο. Είναι η ενημέρωση ω προ τη συνέχιση και των διεκθέσεων, δηλαδή και Goldstone και στο Λίσκου. Και η αποστολή Goldstone και η αποστολή για το Στολίσκο αλλά και η αποστολή της Επιτροπής Συνέχισης της έκθεσης Goldstone, τρεις διαφορετικές αποστολές, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε μεγάλη προθυμία συνεργασίας του Ισραήλ και έγιναν διάφορα διαβήματα. Και αν όντως είχε εκδηλωθεί συνεργασία του Ισραήλ με τις αρμόδιες επιτροπές θα υπήρχε και η προθυμία των επιτροπών ε, να λάβει υπόψη σοβαρά τα σχόλια του Ισραήλ. Αλλά δυστυχώς το Ισραήλ δεν ανταποκρίθηκε στην έκκληση συνεργασίας. Αυτά ήταν τα τελικά συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον Τάρακ Μάρεϊ από το Παλαιστινιακό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχετε το λόγο κύριε Μάρη για 8 λεπτά επίσης. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Θα ήθελα να συνεχίσω και να αναφερθώ στις εσωτερικές έρευνες οι οποίες έγιναν σχετικά με τις συστάσεις Γκόλστον και με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, θέλω να σας πω ποια είναι τα αποτελέσματα μίας έρευνας διότι θεωρώ ότι είναι καλό να έχει κανείς το πλαίσιο αναφοράς όταν κάνει μία εξέταση ε, ε, πρέπει η μελέτη να είναι αποτελεσματική δηλαδή ουσιαστική και να μην είναι για το Θεαθήνε κατά τρόπον ώστε να μπορέσει να ε, εντοπίσει τους υπευθύνους και να οδηγήσει στη δίωξή τους. Επίσης ε, είναι προφανές ότι το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο ο πλήρως χωρίς παρεμβολές από τρίτους. Τρίτη και τέταρτη προϋπόθεση είναι να είναι έγκαιροι ε, και ε, να μπορούν ε, να αντέξουν στην εξέταση από τρίτους και θα σας μιλήσω καταρχήν για τις έρευνες στην Παλαιστίνη και οι ε, κυβερνήσεις στη Γάζα και στη Ραμάλα δημιούργησαν ομάδες οι οποίες ε, θα ε, έκαναν τις έρευνες και δεν μπορούν βέβαια βάσει των προϋποθέσεων να θεωρηθούν ότι είναι εξετάσεις για εγκληματικές ενέργειες διότι δεν έχει γίνει ε, ε, από πλευράς ε, διεθνούς δικαίου μία ουσιαστική πραγματική εξέταση. Και αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι το δίκαιο χρησιμοποιείται μόνο για να δώσει την ψευδέστηση της δικαιοσύνης. Υπάρχουν τρία ουσιαστικά προβλήματα και θα αναφερθώ στο το σύστημα διότι το ε, τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε ε, απορρέουν από πείρα 15 ετίας ε, για τις δικαστικές υποθέσεις. Υπάρχει καταρχήν η προϋπόθεση στην αρχή μίας εξετάσεως ότι οι ε, κανόνες που εφαρμόζονται είναι νόμιμοι ε, και όλες οι διαδικασίες είναι νόμιμες. Ε, δεν γίνεται δηλαδή μία έρευνα παρά μόνο εάν υπάρχουν εξαιρετικές συνθήκες. Δεύτερον, ο μηχανισμός. Υπάρχουν δύο βασικοί μηχανισμοί. Ο πρώτος είναι η επιχείρηση της ενημερώσεως ε, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε investigation on demand το οποίο δημιουργούν ε, οι στρατιωτικοί για να μπορέσουν να διδαχθούν και να δουν πώς οι κινήσεις των στρατιωτικών μπορούν να βελτιωθούν στο μέλλον. Ε, εδώ όμως το πρόβλημα είναι ότι επικαλύπτεται με ε, ε, εγκληματικές έρευνες πράγμα με το οποίο είναι αντικρουόμενο. Είναι ε, ανώνυμα, υπάρχει εξέταση ανωνύμων άρα δεν είναι ουσιαστικό στοιχείο και ένα βασικό στοιχείο όταν ε, εξετάζουμε αυτές τις επιχειρήσεις ε, της ενημερώσεως του debriefing είναι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα απορίσματα σε δικαστήριο διότι αν ε, κανείς τις αμφισβητήσει αμέσως εξαφανίζονται. Προσπαθούμε να αμφισβητήσουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι απτό. Οι δεύτερες μελέτες είναι αυτές οι οποίες γίνονται και οι έρευνες οι οποίες γίνονται από την αστυνομία κατ' εξαίρεση και βασίζονται και πάλι σε αυτές τις ε, ε, επιχειρηματικές ενημερώσεως. Δηλαδή πρόκειται για ε, ένα εξιστήματο, μια εξιστήματος διαδικασία. μεταξύ του 2000 και 2007 Είδαμε ε, ε, 14.000 ε, θύματα που, ε, που είτε ε, σκοτώθηκαν είτε τραυματίστηκαν και ένα ελάχιστο μόνο ποσοστό από αυτές εξετάστηκαν και ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό έφτασε στην απαγγελία κατηγοριών. Μέσα σε 7 έτη Παλαιστινιακό Πρέπει να σας πω επίσης ότι ο Γενικός Εισαγγελέας είναι σύμβουλος εις τους στρατιωτικούς επί θέματα νομοθεσίας και βασίζεται και εις την εφαρμογή του ποινικού κώδικα ε, εκ των υστέρων δε ε, αφού έχει συμμετάσχει στις ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις ελέγχει την κατάσταση ε, για να δει αν πρέπει να απαγγείλει κατηγορίες. Βλέπετε λοιπόν ότι κάποιος πρέπει να εξετάσει την νομιμότητα αποφάσεων οι οποίες εκ προημίου θεωρούνται ε, νόμιμες. Άρα είναι μία ε, τελείως γελία κατάσταση. Σε δύο χρόνια Αχ, στα δύο τελευταία χρόνια έχουν ε, ε, γίνει ε, πολλές έρευνες αλλά κατέληξαν μόνο σε 47 απαγγελίες κατηγοριών. Η οργάνωσή μου είχε υποβάλει 1048 διαμαρτυρίες εκ των οποίων ελάχιστες ένα μικρό κλάσμα μόνο εξετάστηκε σοβαρά και το πρόβλημα με τους εκπροσώπους των θυμάτων ε, είναι ότι δεν ε, γνωρίζουμε τι γίνεται διότι πολλές φορές ε, δεν λαμβάνουμε καμία απάντηση έχουμε λάβει καμιά δεκαριά απλώς απαντήσεις από τους Ισραηλισμούς ένας δύο μόνο καταδικάσεων άρα βλέπουμε ότι είναι μικρό το, το ποσοστό. Ε, δύο στρατιώτες που κατηγορήθηκαν ότι χρησιμοποιούσαν σαν ανθρώπινες ασπίδες ε, πολίτες, ε, παιδιά, απλούστατα είχαν τρεις μήνες κατά τους οποίους δεν μπορούσαν να εξασχίσουν την υπηρεσία τους. Ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο τον Μίρι Βαϊνγκάρντεν, ε, τον ε, ε, Ισραηλινό ακτιβιστή. Την Ισραηλινή ακτιβίστρια, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Προέτους μίλησα εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο επί του αυτού θέματος. Εκπροσωπούσα τρεις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά σήμερα η οργανώσεις αυτές έχουν επιφυλάξεις ε, να εκπροσωπηθούν και να μιλήσουν σε φόρα, <clears throat> διότι έλαβαν ε, κάποιες απειλές, ε, εκποβήθηκαν κλπ. Θα επανέλθω από αυτό τώρα. Σε ό,τι φορά τις έρευνες, να πω ότι οι Ισραηλινές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν συμμετάσχει και σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα ασχολήθηκαν και με την άφηξη των ε, μαρτύρων και καταλήξαμε σε παρόμοια συμπεράσματα με αυτά των κρατικών οργανώσεων σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις ε, που αναφέρθηκαν αλλά και επί ουσίας. δεν ε, υπήρξε καμία απόδοση ευθυνών, δεν υπήρξε λογοδοσία για τα θέματα των ε, παραβιάσεων που όντως υπήρξαν από τον Σεπτέμβριο. Δεν ε, υπήρξαν πολλές νέες εξελίξεις επί της ουσίας. Ξεκίνησε μια έρευνα που έχει είχε διακοπεί σε ό,τι φορά την οικογένεια Σαμούνη Ξέρετε ότι <clears throat> σκοτώθηκαν μέλη αυτής της οικογένειας και δεξάγεται και μια έρευνα σε ανώτατο στρατιωτικό επίπεδο αφορά τον συνταγματάρχη ε, συνταγματάρχη πάνω του Ισραηλινού στρατού. Κάτι ακόμα το οποίο έχει συμβεί από τότε είναι ότι στρατιώτες οι οποίοι συμμετείχαν στην επίθεση ε, έγιναν αντικείμενο ενός δοκιμωτέα μιας ταινίας που γυρίστηκε η έκθεση Goldstone ανέφερε ότι οι επιθέσεις στις ε, μη στρατιωτικές υποδομές ε, έγιναν ε, με πρόθεση <clears throat> και οι στρατιώτες δήλωσαν πως τους δόθηκε εντολή να καταστρέψουν ένα μια εγκατάσταση εκτροφής πουλερικών και αυτό αναφέρεται εξάλλου και στην έκθεση Goldstone και θεωρήθηκε ότι το για εκδίκηση. Όσες περισσότερες προφορίες λοιπόν βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, τότε τόσο περισσότερο θεωρείται ότι τα αναφερόμενα στην έκθεση Γκολστόν είναι αληθή. Και κάτι ακόμα, προτού να μπω στο θέμα των μη κυβερνικών οργανώσεων, από το Σεπτέμβριο συντάχθηκε μια ακόμα έκθεση. Δεν αφορούσε την ε, επίθεση στην ε, Γάζα, και αφορά στην ε, νομιμότητα του αποκλεισμού και η ε, Ερευνητική Επιτροπή κατέληξε στον πέρασμα ότι ο αποκλεισμό είναι νόμιμος και η Επιτροπή Ρόκλ πρόκειται να παρουσιάσει το δεύτερο κομμάτι της έκθεσης λίγο πριν από το Μάρτιο, πριν να ζητηθεί το ζήτημα στην ε, συνέλευση. Και εδώ θίγεται το θέμα της ατιμορρησίας, ε, της ε, έλλειψης λογοδοσίας κλπ. Και τέλος, χθες ένας πρώην στρατιώτης 23 ετών καταδικάστηκε και για διαρροή πληροφοριών σε ό,τι αφορά παραβάσεις, παραβιάσεις μάλλον δικαιωμάτων από τον στρατό και η κεντρική διοίκηση τον καταδίκασε σε δεκαετή κάθεξη. Την περσμένη εβδομάδα υπήρξαν ε, δύο εξελίξεις, ορισμένοι ξυμώνουν να το γνωρίζουν. Ένα ε, αφορά τον ε, νομο, νομοθεσία για την χρηματοδότηση κάποιων οργανώσεων και το άλλο αφορά την κάποιες έρευνες αναφορικά με τις εξαγοράς ε, δημόσιων εκτάσεων. Το νομοθέτημα αυτό πρόκειται να ψηφιστεί στη δεύτερη ανάγνωση και υποθέτουμε ότι η διατύπωση θα τροποποιηθεί. Στην αρχή ήταν πολύ δρακόντια η διατύπωση σιγά σιγά την ε, απάλυναν την διατύπωση αυτού του νομοσχεδίου Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η ψηφοφορία δεν πρόκειται να εξαχθεί αυτή η εβδομάδα που είχε προγραμματιστεί, αλλά την επόμενη. Τώρα, ο νομοσχέδιο αντι-boycott κατά του αποκλεισμού θα ψηφιστεί και <clears throat> αφορά το αποκλεισμό κάποιων ε, προϊόντων ε, αρχικά και εδώ η διατύπωση ήταν πολύ σκληρή και μια που έχει τελειώσει ο χρόνος μου είμαι στη για περαιτέρω απαντήσεις σε σχόλια σας. Ευχαριστώ κυρία Βαϊγκάρντεν. Πολύ θετικές αυτές οι ειδήσει για όσους ε, παρακολουθήσαμε αυτή την περίπτωση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και... Στο Ισραήλ, που υποτίθεται είναι δημοκρατική χώρα, ε, εφαρμόστηκαν τέτοια δρακόντια μέτρα και μάλιστα εκστρατεία εκφοβισμού κατά ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι αβάσιμες κατηγορίες, τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι αντάξεις ε, απολυταρχικών καθεστώτων σαν αυτών της Τινησίας, όχι μιας δημοκρατικής χώρας όπως είναι το Ισραήλ. Θα δώσω τώρα το λόγο στα μέλη της Υποεπιτροπής, πρώτα στην κυρία Άουγκεν. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και για τις εισηγήσεις σας. Δυστυχώς οι πληροφορίες αυτές μας αφήνουν άναυδους, όπως πάντα είναι συγκλονιστικές αυτές οι ειδήσει και παρόλο που υπάρχουν κάποιες ε, μικρές βελτιώσεις, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι τραγική και γίνεται όλο και πιο αναξιόπιστη αυτή η θέση ότι το Ισραήλ είναι από τις χώρες τις οποίες μπορούμε να βασιστούμε γιατί πραγματικά έπιασε πάτο, έφτασε στο να σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό από πολλές απόψεις σε πολλές περιπτώσεις έχουμε μια ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις Γενέβης όταν πραγματεύεται αυτά τα θέματα. Δεν θα πρέπει στη συνέχεια να δούμε μια διχασμένη Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς σαφή και διατρανωμένη θέση, γιατί έτσι θα χάσουμε πάσα αξιοπιστία. Έχω μια ερώτηση κάπως δύσκολη πήγαμε μια αντιπροσωπεία για την Παλαιστίνη πρόσφατα στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη και μάλιστα όταν βρεθήκαμε στη Γάζα ακούσαμε από ανεπίσημες πηγές ότι η Χαμάς βλακοδός είχε ουσιαστικά υιοθετήσει αυτή την ιδέα της ε, δολοφονίας αμάχου πληθυσμού και μάλιστα βλέπαμε ε, αφήσει στους δρόμους της Γάζας που έλεγαν ότι αυτοί οι άνθρωποι που φαινόταν στις αφήσει ε, ήταν άνθρωποι που τους σκότωσαν ε, στο κρεβάτι στον ύπνο τους μέλη του άμαχου πληθυσμού. Ήταν πραγματικά ανόητο ότι η δράση της Χαμάς ουσιαστικά ε, ανέδειξε σε μάρτυρες, ανέδειξε σε μάρτυρες αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε τίποτα για αυτή την εκστρατεία. Γιατί από ό,τι άκουσα ήταν γνωστή αυτή η περίπτωση στη Γάζα, ότι οι Χαμάς και οι άλλοι βρήκαν τις αρεσκίες τους αυτή την θέση. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω κάποιες πληροφορίες, αν γνωρίζετε το περιστατικό και πώς έγινε τι έγινε στον πόλεμο της Γάζας, πώς ήταν οι άμαχοι που έχασαν τη ζωή τους. Έγινε σωστή καταμέτρηση των θυμάτων. Πραγματικά με κατέπληξε αυτή η πληροφορία και δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποια στοιχεία για να μας ενημερώσετε. Ευχαριστούμε κυρία Άουγκεν. Δεν ζήτησε άλλος κανείς το λόγο. Α, η κυρία Κιλ Νίλσεν. Σας ευχαριστώ. Αυτά που ακούσαμε είναι αρκετά αποκαρδιωτικά αλλά δεν μας εκπλήσουν γιατί χρόνια ολόκληρα έχουμε μια συνενοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενισχύει αυτό το δικαίωμα, αυτό το δίκαιο της ατιμορρησίας και αυτή την αίσθηση ότι θα παραμείνω ατιμόρυτη ή ένοχη. Και η κυβέρνηση αυτή που είναι ε, ακροδεξιά κυβέρνηση και θα πρέπει να λέμε τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη και τα πράγματα με το όνομά τους ουσιαστικά ακυρώνει οποιαδήποτε προσπάθειά μας για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη μας στον Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε για το, την κατάσταση στο Ισραήλ. Είχαμε συναντήσεις και δημόσιες ακροάσεις και με μη κυβερνητικές οργανώσεις και καταδικάσαμε αυτή την παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης και την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ισραήλ. Καταδικάσαμε το, τον αποκλεισμό της Γάζας, μιλήσαμε για την έκθεση Goldstone, πρόσφατα πήγαμε στη Γάζα και μάλιστα εγώ μέσα σε ένα εξάμεινο πήγα δύο φορές στη Γάζα και διαπιστώνουμε ότι στη Γάζα έχουμε όλο και περισσότερα παιδιά που λιμοκτονούν που υποσυντίζονται η Ούνρα δεν μπορεί να ε, εξασφαλίσει τρόφιμα σε αυτά τα παιδιά δεν μπορούν αυτά τα παιδιά να φοιτήσουν στο σχολείο γιατί τα σχολεία τους βομβαρδίστηκαν και αυτό είναι γεγονός, το είδαμε με τα μάτια μας και μάλιστα το αναφέρει και η έκθεση Κολστών. αλλά δεν, χρειάζεται καν, δεν χρειαζόμαστε καν την έκθεση Κολστών, αρκεί κανείς να πάει στη Γάζα και να, να δει ότι τα ε, σχολεία έχουν καταστραφεί από βομβαρδισμό και δεν μπορούν να, να, ε, να κατασκευαστούν γιατί απαγορεύεται η εισαγωγή δομικών υλικών για την ανέγερση αυτών των σχολείων. Με τον αποκλεισμό ήταν ε, τεράστιες ε, οι αλέθρες συνέπειες και είναι πραγματικά σκανδαλός που δεν δόθηκε καμία συνέχεια μετά την έκθεση Goldstone. Η έκθεση Goldstone αναφέρθηκε στην πιθανότητα προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ελήψη ε, αξιόπιστης έρευνας μέσα σε ένα εξάμεινο. Και εκεί βρισκόμαστε. Εντός εξαμήνου δεν έγινε καμία αξιόπιστη έρευνα τι περιμένει λοιπόν ο ΙΕ για να προσφύγει στο Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Θα πρέπει επιτέλου να δράσουμε τέρμα τα λόγια, τέρμα οι εκθέσει. Αρκετό χρόνο χάσαμε με τα λόγια και τι εκθέσει. Εμεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, ω Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει κατεπηγόντω να αναλάβουμε δράση. Πριν από λίγο μιλήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο η στρατιωτική ε, ε από στρατιωτική σκοπιά το θέμα της νεοπομπής θα πρέπει να δούμε τι έγινε και από πλευρά άμαχου πληθυσμού ή πολιτών. Ε, μια νέα ευρωπαϊκή νεοπομπή ετοιμάζεται και ξέρω ότι στην ε, Γαλλία γίνονται τακτικά συναντήσεις και σε πολλές χώρες Ευρώπης υπάρχει ε, κινητοποίηση, γίνονται έρανοι για συλλογή χρημάτων και έχουν που ετοιμάζονται και στρατιωτικών που θα συμμετέχουν στην Ιωπομπή. Θα έχουμε και βουλευτές που θα συμμετέχουν σε αυτή την υπομπή. Ελπίζω να μην ε, έχουμε την ίδια κατάληξη με τον προηγούμενο στο Λίσκο και με θύματα. Ετοιμάζεται λοιπόν αυτή, αυτή η νέα νιοπομπή για να καταγγείλει την, τον αποκλεισμό. Πολίτες ε, κινητοποιούνται για να συγκεντρώσουν τα χρήματα γιατί είναι πολύ δαπανηρή αυτή η διαδικασία. Οι πολίτες λοιπόν κάνουν το έργο τους, αλλά δεν ε, τους συνοδεύουν οι πολιτικοί με αντίστοιχε πρωτοβουλίες. Οι πολίτες πάλι αναλαμβάνουν τους κινδύνους ε, και καταγγέλουν αυτή την, αυτό το σκανδαλώδη αποκλεισμό της Γάζας. Δεν υπάρχει όμως καμία αντίστοιχη υποστήριξη από τους πολιτικούς. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε, αν μη τι άλλο για την ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί ακόμη και οι μερίδες του φαγητού είναι ανεπαρκείς. Κάτι που με συγκλώνησε το Μάιο είναι ότι τα παιδιά της Γάζας δεν έχουν καν παπούτσια. Τις περισσότερες φορές κυκλοφορούν ξυπόλυτα και πραγματικά υπάρχει επιδείνωση σχέση με την προηγούμενη φορά. Τα παιδιά κυκλοφορούν ξυπόλυτα παντού. Μέσα στα μπάζα από τα καταδαθισμένα σπίτια από το βομβαρδισμό. Και κανένα φαίνεται να μην ενισχύει. Λέμε υπάρχει αποκλεισμό στην Γάζα. Και τι έγινε. Θα πρέπει να καταδικάσουμε αυτή την σκανδαλώδη πραγματικά και φρικα, φρικαλέα κατάσταση. Αρκετά είπαμε τους τελευταίους μήνες. Οι συνέπειες αυτής της επίθεσης εκ μέρους του Ισραήλ είναι ορατές όταν πηγαίνει κανείς επί τόπου. Βέβαια τους νεκρούς δεν τους βλέπουμε, ακούσαμε ότι υπάρχουν θύματα, ακούσαμε για νεκρούς, υπάρχουν οι αφήσει, αλλά τους τραυματίες τους βλέπουμε. Υπάρχουν και τραυματίες, πολλοί άριθμοι είναι οι τραυματίες στη Γάζα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολύ μήνυ έρευνα για να δούμε τι συνέβη. Γνωρίζουμε τα γεγονότα. Ας αφήσουμε λοιπόν τις υποκρισίες. Και τέλος θέλω να πω ότι ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Ναβί Πίλε, πήγε την Κυριακή το απόγευμα στο Ισραήλ για την πρώτη επίσκεψη στα Παλαιστινιακά εδάφη και στο Ισραήλ και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις του Ισραήλ και της Παλαιστίνης καλωσόρισαν την άφηξη της ύπατης και μίλησαν και ζήτησαν μάλλον την εφαρμογή της ε, έκθεσης Goldstone. Αυτά ακούσαμε ε, την ε, Κυριακή. Υπάρχει αυτή η έκθεση, είναι σοβαρή, θα πρέπει λοιπόν επιτέλους ε, να την εφαρμόσουμε. Αυτά. Δεν έχω καν ερώτηση, αλλά έπρεπε να πω κάτι. Ευχαριστώ. Τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον υπο... αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, ακούσαμε τους φιλοξενούμενους μας και ακούσαμε την κυρία Κιλ Νίλσεν και άλλους, ε, την κυρία Άικεν και ε, αυτό επιβεβαιώνει αυτό το οποίο σκεφτόμουν. Ότι δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να υπεραμεινθούμε των ε, αξιών μας, των αξιών ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ιδίως ε, όταν πρόκειται για κράτη με τα οποία έχουμε μακροχρόνιες σχέσεις τα ανθρώπινα δικαιώματα φαίνονται να βρίσκονται ε, σε ε, πιο, ε, να μην αποτελούν προτεραιότητα και αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι παραπάνω εκθέσεις και αποστολές οι οποίες επιβεβαιώνουν συνήθως αυτά τα οποία ήδη γνωρίζουμε. Δηλαδή είναι σαφές ότι υπάρχουν σοβαλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπάρχουν ορισμένοι μηχανισμοί ε, διεθνούς δικαίου που μας επιτρέπουν να επιλύουμε τις περιπτώσεις τέτοιων παραβιάσεων και πρέπει να επιζητήσουμε κάποιο αποτέλεσμα το ταχύτερο δυνατόν. Σαν ευρωβουλευτές θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ακριβώ το χαρακτηριστικό και να εξετάσουμε διάφορες εκθέσεις που αναφέρονται στις σχέσεις μας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Ισραήλ, Ισραήλ διότι επί του θέματος αυτού ε, δεν υπάρχει και μεγάλη κινητικότητα. Το πιο βασικό το οποίο μπορώ να πω και το οποίο ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε μία ηθική ευθύνη και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να ε, κλείνουμε τα μάτια σε τέτοιες καταστάσεις. Ακόμη και αν δεν είναι πολύ βέβαιο ποιο θα είναι το μέλλον της εκθέσεως Goldstone, και ακόμη και αν ε, δεν ε, ε, υιοθετηθούν όλες οι συστάσεις παρόλα αυτά έχουμε ευθύνη και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ρωτήσω τους φιλοξενούμενους μας πώς ακριβώς φαντάζονται ότι μπορούν να ερμηνευθούν σε συγκεκριμένα μέτρα αυτές οι συστάσεις. Θα πρέπει τώρα να ζητήσουμε από τον κύριο Μαρσέλο Φαράτζη να λάβει τον λόγο συντομία διότι είναι ένας γνωστός δημοσιογράφος ο οποίος είναι εδώ, παρακολουθεί τη συζήτησή μας και πιστεύω ότι για ένα-δύο λεφτά Καλό θα ήταν να μας πείτε ε, τα, τις εμπειρίες σας σαν αυτόπτη μάρτυρα και μετά θα ζητήσουμε από την, ε, από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσεως να ε, αντιδράσει και για να σχολιάσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε Επί 20 χρόνια ήμουν απεσταλμένος στις Βρυξέλλες και σαν ανταποκριτής για την οργανωμένη ε, την οργανωμένη εγκληματικότητα αλλά ποτέ δεν φοβήθηκα τόσο πολύ όσο, όσο ε, πρέπει να παρουσιάσει την έκθεσή για το σκολί, στο Λίσκο και τώρα υπάρχουν ένα-δυο γεγονότα τα οποία είναι λίγο πολύ γνωστά. Μιλάμε για ένα πλοίο ενώ φαίνεται ότι ο στόχος ήταν να πούμε ε, στο κοινό ότι μόνο μία χώρα είχε εμπλακεί, η Τουρκία. Δεν όμως αυτό το οποίο εγώ διεπίστωσα όταν ε, είχα πάει υπήρχαν δύο πλοία, 37 ε, εθνικότητες από όλο τον κόσμο και αυτό που δεν ελέγχθη στο κοινό ήταν ότι ε, ότι δεν υπήρχε επίθεση μόνο εναντίον του πλοίου και των ε, ε, ανθρώπων αλλά εναντίον των ε, μέσων ενημέρωσης και του εξοπλισμού μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σούλ, τον κύριο Ντόλ, τον κύριο Φερχόφστατ Κονβεντίτ από την διάσκεψη των Προέδρων που ζήτησαν από τον Πρόεδρο Μπούζεκ να ε, ε, ε, γράψουν στις Ισραηλινές αρχές που κατάσχεσαν τον εξοπλισμό μας. Εγώ δεν έχω καταφέρει να πάρω πίσω τίποτα και αυτό είναι μια άλλη πραγματικότητα. Άκουσα λοιπόν ότι εσείς εδώ είσαστε στενά συνδεδεμένοι με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία του τύπου που είναι μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να πούμε ολόκληρη την αλήθεια γιατί είχαμε κρύψει ορισμένα τμήματα της ανταποκρίσεως και ετοιμάζουμε τώρα μετά από ένα χρόνο δηλαδή στο τέλος Μαΐου εφέτος ένα ντοκιμοντέρ όπου θα δείτε ορισμένες πληροφορίες στο διαδίκτυο επ' αυτού και ε, αν ε, ε, βάλετε βι info θα το βρείτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για αυτές τις πληροφορίες και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Τογιώνα από την, εξωτερική την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ. Είμαι ευγνώμων για τις παρουσιάσεις ε, που έφτασαν εγκαίρως. Σε ό,τι αφορά την έκθεση Goldstone, εμείς ε, ζητήσαμε από όλες τις ε, τους να ξεκινήσουν ανεξάρτητες ε, έρευνες σε ό,τι αφορά την παραβίαση των διεθνών κανόνων και του διεθνούς δικαίου. Εμείς συνεχίζουμε να θίγουμε το ζήτημα αυτό και σε διμέρες επίπεδο. Μετά από την έκθεση της Επιτροπής των Πυρογνωμόνων του Σεπτεμβρίου, με βάση λοιπόν τα ευρήματα θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες και από τις αρχές του Ισραήλ αλλά και από τις αρχές της Παλαιστινιακής για προκειμένου να εφαρμοστεί η αρχή της λογοδοσίας. και να εξετάσουν τις παραβιάσεις, τις παραβιάσεις. Φυσικά και προσβλέπουμε στην ε, έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που θα την παρουσιάσουν στις, ε, στο εγγύς μέλλον και για την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης ε, αυτό που έχει σημασία είναι να παραμείνει ενωμένη και να στείλει ένα μήνυμα προς τους εμπλεκόμενους Την τελευταία στιγμή όμως ε, υπήρξαν και άλλες εκθέσεις ε, πέραν της ε, εκθέσεως Goldsmith όπως γνωρίζετε Για το στις 15 ήμασταν καλά προετοιμασμένοι τώρα προετοιμασμόστε για το έτσι 16 Τώρα, σε φορά την ε, ζήτημα του Στολίσκου και την σχετική έρευνα, θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει συντονισμό ε, και τη Ανεξάρτητης Επιτροπής αλλά και της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, το Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που ανέκρινε την έκθεση για το θέμα αυτό είδαμε ότι υπήρχαν κάποιες ε, ελλείψεις ε, σε αυτήν τις οποίες προσπαθούσαμε να, προσπαθούσαμε να καλύψουμε με, στην προσεχή έκθεση που θα υποβάλουμε. Φυσικά βλέπουμε ότι η ετοιμότητα και των ε, Παλαιστινιακών χωρών και του Ισραήλ να συνεργαστούν με τον Γενικό Γραμματέα και ελπίζουμε ότι τα συμπεράσματα θα μπορέσουν να παρουσιαστούν συντόμως. Τώρα για την κατάσταση στην Γάζα συμφωνούμε με τις ε, ανησυχίες που εκφράστηκαν και ζητάμε την ε, ανεφόρον ξεκίνηση διαπραγματεύσεων και την άρση του αποκλεισμού. Θεωρούμε λοιπόν θετικό στοιχείο να επιτρέψει η κυβέρνηση κάποιες ε, εξαγωγές. Χρειάζεται να υπάρξει ένα <clears throat> συνεκτικό πακέτο για Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά την παροχή ανθρωπικής βοήθειας, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασικός ε, εμπλεκόμενος, όπως και η υπηρεσία έργων των ΗΕ. Ευχαριστώ κύριε Τόιρμαν. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Άουγκεν και μετά στην κυρία Βάν Γκάρδεν και στην κυρία Μάρη για να απαντήσουν. Αλλά και στην κυρία Άρβιτσον. Κυρία Άουγκεν. Εν συντομία, μία Ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Αν, αν είναι η Τσεχία ή η Ολλανδία να αποφασίσουν ποια είναι η θέση τους, καλύτερα να έχουμε μια σαφή θέση παρά τη, τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Να σας πω τι είδαμε στη Γάζα με τα, την ακρόαση και με την ύπατη αρμοστία. Δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση με το άνοιγμα των, των περασμάτων. Και μάλλον πρόβλημα δημιουργήθηκε παρά α, λύση σχεδόν απαγορεύεται απόλυτα η εισαγωγή δομικών υλικών στη Γάζα. Και αν δεν ε, επιτρέπεται η εισαγωγή δομικών υλικών, πώς θα αναπτυχθεί η Γάζα. Η Γάζα τελεί ε, υποπολιορκία. Έχουμε συνέχεια στρατεύματα και αυτό είναι παράνομο. Επίσης η κατάσταση στα περάσματα είναι ακόμη χειρότερη γιατί το Ισραήλ κλείνει όλα τα περάσματα με εξαίρεση το Καρέμ Σαλόμ. Όλα θα πρέπει να καταβαίνουν εκεί για να περνάνε. Και καθημερινά στη Γάζα σκοτώνονται παιδιά Και η κατάσταση και για την υπατηρμοστία είναι δύσκολη γιατί είναι πολύ δαπανηρή η διαδικασία και όλα περνάνε μέσα από ένα στενό διάδρομο που ένα και μόνο πέρασμα που έχει παραμείνει ανοιχτό. Μα λένε ότι έχει βελτιωθεί κάπω η κατάσταση, αλλά σα διαβεβαιώ ότι είναι αναλυθέ αυτό και ανακριβέ. Έχουμε βαρεθεί να ξανακούμε τα ίδια και τα ίδια υποτίθεται από ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση. Now, um... Ευχαριστούμε κύριε Άουγκεν. Η κυρία μετά από αυτά που είπε η Μάργαρετ Άουκερ που μίλησε για το κουαρτέτο. Το κουαρτέτο θα συνεδριάσει το Σαββατοκύριακο. Α, πλήρης αποτυχία, καμία επίσημη δήλωση, παταγώδης αποτυχία το κουαρτέτο, έχει γελιοποιηθεί πλήρως το κουαρτέτο και αυτό διασκεδάζει τους Ισραηλινούς γιατί τους συμβουλεύουν να ε, εγκαταλείψουν τις ερευνευτικές διαδικασίες και να επικεντρωθούν στην καταπολέμηση της φτώχειας στη Μέση Ανατολή. Έγιναν πολλές ηρωνικές δηλώσεις ε, εκ μέρους Ιραηλινών για το κουαρτέτο. Το κουαρτέτο πραγματικά είναι μια καταστροφή. Δεν έχει λύσει τίποτα στο πρόβλημα, μάλλον αποτελεί τμήμα του προβλήματος στο κουαρτέτο. Ευχαριστούμε κύριε Νίλσεν. Ε, Ο κύριος Μάρη, ως προς το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ε, καταλήξει σε δύο χαρακτηριστικά της ε, ε, της κατάστασης, η ατιμορρησία και η κλιμάκωση της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι τα δύο αυτά βασικά χαρακτηριστικά. Γίνονται υποτίθεται έρευνες, αλλά δεν αποδίδεται καμία δικαιοσύνη, δεν αποδίδεται καμία κατηγορία και δεν απονέμεται καθόλου δικαιοσύνη. Γίνονται εχώριες υποτίθεται έρευνες που επίσης απέτυχαν με βάση τις συστάσεις της έκθεσης Goldstone, αλλά και με τις απαιτήσει του διεθνούς δικαίου, η κατάσταση θα πρέπει να μεταφερθεί τώρα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Πρέπει να γίνει προσφυγή εκεί. Η διαδικασία Goldstone πέρασε από τη Γενέβη στη Νέα Υόρκη και από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει να γίνει ε, να διεξαχθούν πια διεθνείς έρευνες και να απαγγελθούν διεθνώς κατηγορίες. Και αυτό είναι ένα από τα θεμέλια των βασικών αρχών που αναφέραμε προηγουμένως. Για το κουαρτέτο τώρα και είναι η βασική θέση και της είπα της αρμοστίας. Το πρόβλημα είναι να γίνει μια θεσμοποίηση αυτής της κατάστασης. Μιλήσα, μιλήσαμε για μερική, μερικό αποκλεισμό ή μερική απελευθέρωση. Το θέμα είναι ότι μισό εκατομμύριο άνθρωποι τιμωρούνται καθημερινά και ο κίνδυνος είναι να νομοποιηθεί αυτή η κατάσταση με τη συνενοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί θα πρέπει να είμαστε πολύ κατηγορηματικοί. Αυτά και να δώσω το λόγο στη συνάδελφο. Σας ευχαριστώ για την σαφή αυτή δήλωση. Κύριε Βάινκαρτ. Σχετικά με το τι μπορεί να γίνει Ξέρετε, γνωρίζετε τα μέσα, τα εργαλεία καλύτερα από ότι εμείς, αλλά υπήρξε ένα ψήφισμα στο Κοινοβούλιο και θα μπορούσαμε να ζητήσουμε απαντήσεις από την είπα την εκπρόσωπο κυρία Άστον αναφορικά με την πρόοδο, την την εφαρμογή αυτού του ψηφίσματος. Στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου θα πρέπει να εξετάσουν το θέμα αυτό αλλά και σε διάφορα φόρα όπως Ευρωπαϊκή Ένωση Ισραήλ στο Συμβούλιο το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε αυτή τη συνάντηση του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ αλλά και το ζήτημα της ατιμορρησίας. Προέτους, όπως σας είπα, σας είχα ξαναπεί περίπου τα ίδια πράγματα. Δεν έχει υπάρξει πρόοδος στο Ισραήλ επί του θέματος. Αυτό που είδαμε είναι ότι στις ψηφοφορίες τόσο στη Γενέβη όσο και στη Νέα Υόρκη υπήρξε κάποια σύγχυση. σε ό,τι αφορά τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 50 κρατη λοιπόν δεν ε, συμφωνούν μεταξύ τους και άρα δεν μπορεί να υπάρχει μια συμπεφωνημένη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε θα πρέπει να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Ευχαριστώ κύριε Άρβινσον. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα, όπως είπε ε, η κυρία Νίλσεν, ότι εκπρόσωπος βρίσκεται τώρα στα κατεχόμενα. Uh, και συνάντησε τον ε, Σίμων Πέρες ε, και τους ε, αρμόδιους από την Παλαιστινική Αρχή. Το θέμα της λογοδοσίας τόσο η κυρία Άστον όσο και ο Γενικός Γραμματέας επιμένουν ε, περί της λογοδοσίας ε, όπως επίσης ε, επιμένουν και για το ζήτημα του αποκλεισμού και καλούν την άρση του αποκλεισμού και την άρση της ατιμορρησίας επίσης πολλές μη κυβερνικές οργανώσεις αλλά και άτομα τα οποία συμμετείχαν στην ε, σύνταξη του ε, κόρθων και στην συνεργασία ε, έχουν γίνει αντικείμενα απειλών. Αυτά. Ευχαριστώ. Να επαναλάβω ότι έχει ήδη πει το Κοινοβούλιο. Καλεί την εφαρμογή της ε, έκθεσης ε, το ζήτημα της ε, λογοδοσίας για θέματα παραβιάσεων επίσης και η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι ο χώρος τον οποίο θα πρέπει να φροντίσουμε να προωθηθεί το ζήτημα της λογοδοσίας και της ατιμορρησίας. και να πρωτοστατήσουμε ομού με το κοινοβούλιο στο σύνολό του. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω αυτό το σημείο της διατάξεως θέμα που είναι ύψη τη σημασίας για την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τώρα το επόμενο σημείο είναι πολύ σύντομο. Σημείο 6. Και εδώ στο λόγο στον Αντιπρόεδρο κύριο Ξύπ. Να σας πω ότι σύμφωνα με τα όσα προείπαμε στην 16η Σύνοδος ε, από 28 Φεβρουαρίου έως 26 Μαρτίου θα διεξαχθεί η σύνοδος στη Γενέβη, θα στείλουμε μια αποστολή και υπενθυμίζω ότι η Γραμματεία θα πρέπει να ενημερωθεί αναφορικά με τους δύο ορισμούς των μελών σε αυτή την αντιπροσωπεία και η καταληκτική προθεσμία είναι αύριο το μεσημέρι 12.00 για την υποβολή υποψηφιότητων με την γραπτή διαδικασία είχε αποφασιστεί ότι θα καταρθεί ψήφισμα το οποίο θα θέτει τις ε, προτεραιότητες και τις ε, θέσεις μας ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ειδικά τα θέματα της αναθεώρησης ε, που μας απασχόλησαν νωρίτερα. Οι πολιτικές ομάδες λοιπόν θα υποβάλουν ένα σχέδιο ψηφίσματος η οποία και θα ολοκληρώσει τη συζήτηση που θα ακολουθήσει μετά από δήλωση της Αντιπροέδρου και είπα της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρία Άστον. Το ψήφισμα λοιπόν θα αποτελέσει και την νομική βάση για περαιτέρω αποφάσεις. Ωραία. Δίνω λοιπόν την Προεδρία στον κύριο Ξύμπ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Περνάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο πρέσβη Έγκελμπερ Τόιερμαν, πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόκειται για ένα στοιχείο της νέας δομής που δημιουργήθηκε μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριος Πρέσβης είναι σημαντικός αξιωματούχος σε αυτή τη νέα δομή και σας ευχαριστούμε θερμά γιατί ε, ως αυστριακός διπλωμάτης είχατε πολύχρονη εμπειρία και θα εμπλουτίσετε με τις γνώσεις σας ε, το Συμβούλιο, την Ειδική Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα σημείο που βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής της δικής μας υποεπιτροπής. Εμείς ως Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τη συνεργασία με την Ειδική Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου και μας ενδιαφέρει η ενεργός δραστηριοποίηση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, τήρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω το λόγο για να ακούσουμε την ομιλία σας, γιατί όπως σας είπα αναγνωρίζουμε τη θέση της ΚΟΧΟΜ, της ειδική Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ως ακρογωνία ολίθου της νέας αρχιτεκτονικής που δημιουργείται με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έχετε 10 λεπτά με βάση το χρόνο που δίνουμε στους προσκεκλημένους μας για να μας ε, παρουσιάσετε την ομιλία σας. Um, σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε και ευχαριστώ την κυρία Χάουταλα την πρόεδρο που με προσκάλεσε στη συνεδρίαση τόσο νωρί μετά την ανάληψη των νέων μου καθηκόντων. Όπω σα είπα, έρχομαι ενώπιον σα ω πρώτο αντιπρόεδρο τη ΚΟΧΟΜ μετά τι νέε ρυθμίσει τη συνθήκη Λισαβόνα και υπό την ε, αιγίδα τη ΥΠΑ τη ε, εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική. Βέβαια, ε, αναφέροντα το ρόλο του Προέδρου της ΚΟΧΟΜ, φαίνεται ότι είναι μια βραχυχρόνια δραστηριότητα. Αλλά σίγουρα το νέο σύστημα είναι πολύ πιο βελτιωμένο από το προηγούμενο που ήταν εξάμεινη διάρκεια. Έτσι εξασφαλίζεται μεγαλύτερη συνοχή, συνέπεια, αλλά δημιουργεί και περισσότερες προκλήσεις. Την πρόκληση της άμεσης ε, μετάβασης που αντιλαμβάνω, και εγώ ως πρόεδρος Κοχόμ αλλά η διαδικασία είναι έντονη γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ σημαντικός ε, τομέας και το θέμα είναι να κρατήσουμε την ενεργό συμμετοχή των 27 χωρών σε θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και ιδιαίτερα σε θέματα πολιτικής ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων. Στο παλιό σύστημα της Προεδρίας είχαμε τον πρόεδρο της Κοχόμ που ταυτόχρονα ήταν και ε, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αναλάμβανε όλα τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με το νέο σύστημα, ο ρόλος του Πρόεδρου της ΚΟΧΟΜ είναι πιο περιορισμένος και παρουσιάζεται ως εξής ο ρόλος αυτός. Η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και σωστής διαχείρισης ΚΟΧΟΜ και εξασφάλιση της λήψη υπόψη της ομάδας των 27 χωρών στη διαμόρφωση πολιτικής στην, εξωτερική στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εξωτερική δράση. Είναι διαφορετικός λοιπόν ο ρόλο του νέου πρόεδρου της ΚΟΧΟΜ σε σχέση με το καθεστώς που ίσχυε προηγουμένω. Οι λεπτομέρειε των ευθυνών και αρμοδιοτήτων μου θα πρέπει να τύχουν αντικείμενο τακτική επεξεργασία ε, και να αξιολογηθούν σε ένα ευρύτερο χρονικό διάστημα. Βέβαια, η προσπάθεια που καταβάλουμε είναι ομαδική προσπάθεια και στην ΚΟΧΟΜ και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βερονίκα Νό είναι η προϊσταμένη για, για τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ανέλαβε δέσμευση να λειτουργήσει πλήρως αυτή η διεύθυνση και αυτό θα φανεί και στην έκθεση πρόοδου με την πρόταση της συγχώνευσης των δύο μονάδων ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γραμματείας του Συμβουλίου, όπως φαίνεται στο νέο οργανόγραμμα που προτείνουμε. Σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη, ο ρόλος μου είναι να φέρω τις ε, θέσεις τους επιτάπητος και να λαμβάνονται αυτές οι υπόψεις στη διαμόρφωση της πολιτικής. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ενεργό ανάμειξη των κρατών μελών στην διαμόρφωση αλλά και στην εκτέλεση της πολιτικής και στις Βρυξέλλες αλλά και σε διμερή και πολυμερή φόρα. Χρειαζόμαστε και πολιτική συμμετοχή και τεχνική υποστήριξη από τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε μια ισχυρή και αξιόπιστη φωνή. Θα πρέπει φυσικά να, να ενισχύσουμε το σύστημα των ομάδων κρούς, ομάδων εργασίας και αυτό θα φανεί στην επόμενη ε, συνεδρίες όπου θα στηθούν νέες ομάδες εργασίας για τους ομοφιλοφίλους, διαφιλικούς κτλ. και την ε, ελευθερία θρησκευτικής πεποίθησης. Είναι σημαντική συνεργασία μας επίσης με την Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουμε δεσμευτεί για στενή συνεργασία με την υποεπιτροπή σα και είμαστε στη διάθεσή σα να ερχόμαστε για ανταλλαγή απόψεων όποτε μα το ζητήσετε και θα λάβουμε υπόψη και τι δικέ απόψει στο έργο μα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τι προσπάθειε και των ΜΕΝ και των ΔΕ για την προώθηση και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διεθνώ. Θα συνεχίσουμε φυσικά τη συνεργασία μαζί σα και ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα και η Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή ε, και η ίδια η πρόεδρος της Επιτροπής θα έρθει να εκφωνήσει ομιλία στην ΚΟΧΟΜ. Σα θεωρούμε έναν πολύ απαραίτητο εταίρο μας και θέλουμε να το υπογραμμίσουμε αυτό. Σε ό,τι αφορά το έργο της ΚΟΧΟΜ για το 2011, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα ειδικά ζητήματα. Ιδίως σε αυτή τη μεταβατική πολιτική ε, περίοδο το πιο ουσιαστικό είναι να μπορούμε να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την ε, ε, το πρόγραμμα των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, σε, και των διαφόρων πτυχών του, δηλαδή διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή στη Γενέβη ή στη Νέα Υόρκη και σε άλλα μέρη και στο Στρασβούργο βέβαια. Επίσης το ΚΟΧΟΜ, δηλαδή το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πέρυσι ε, κατήρτισε ένα πρόγραμμα και ε, στρατηγικές καταχώρες ε, για τις αντιπροσωπείες που βρίσκονται επί τόπου και που θα ακολουθήσουν και άλλα θέματα. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την δεδομένη κατάσταση στη συγκεκριμένη χώρα θα μπορεί να υπάρξει μία πιο σαφής εφαρμογή και μία καλύτερη ένταξη της, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άλλα σημεία. Ο Μισελ Τίλεμανς κατά την Βελγική ε, Προεδρία ε, υπέβαλε ένα, πρόγραμμα ε, και σε συνεργασία με το Συμβούλιο ε, για την Μπρουζ ε, όπου είχαν υποβληθεί πολλές προτάσεις για την ύπατη εκπρόσωπο. Ε, και ε, αυτά πετέλεσαν και την βάση της δηλώσεως ε, πέρυσι στις 15 Δεκεμβρίου όταν συζητήθηκε η συζήτηση και δεσμεύτηκε η εκπρόσωπος υπάρχουν ε, υπεύθυνοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διάφορες αντιπροσωπείες ε, ε, διεθνώς. Το βασικό θέμα για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ότι θα πρέπει να προωθηθεί αυτή η διαδικασία αφού συζητηθεί εσωτερικά κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τα απορίσματα στα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στα κοινοβούλια. Επίσης υπάρχουν και άλλες ε, καινούργιες μέθοδοι εργασίας του Συμβουλίου, ιδίω πρέπει να υπάρχει μία μορφή με μία βάση στο, στις δεν υπάρχει ομοφωνία για μια τέτοια κίνηση και θα χρειαστεί ακόμη χρόνος ε, για να το συζητήσουμε και να κάνουμε και επιπλέον προσπάθειες για να βελτιώσουμε ε, το κοχόμ για να μπορέσουν οι συζητήσεις να γίνουν πιο ουσιαστικές και να έχουμε καλύτερη προετοιμασία κατά τρόπον ώστε να υπάρχουν πιο συγκεκριμένες συζητήσεις. Άρα προς το παρόν το κοχόμ θα συνεχίσει τις ε, μηνιαίες συναντήσεις μια μισή μέρας και θα συγκαλούνται και έκτακτες συνεδριάσεις ε, ε, όποτε αυτό χρειάζεται κατά τρόπον ώστε να καταρτιστούν παραδείγματο χάρη οι στρατηγικές κατά χώραν ε, του Συμβουλίου έχουμε το, την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου μία συνεδρίαση είχαμε ήδη μία και τέλος Φεβρουαρίου θα υπάρξει μία τρίτη άρα βλέπετε ότι εντείνεται η ε, συχνότητα των συνεδριάσεων όποτε χρειάζεται. Αλλά ουσιαστικά οι συνεδριάσεις πρέπει να γίνεται, ε, ε, θα πρέπει να γίνονται στις Βρυξέλλες και να υπάρχουν κατάλληλες εστιασμένες συνεδριάσεις πρώτων μεγαλύτερων συζητήσεων για να μπορούν οι μόνιμες αντιπροσωπείες στις Βρυξέλλες που εμπλέκονται περισσότερο στην εργασία του Συμβουλίου να συμβάλλουν στην καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος του Συμβουλίου. Βάσει ε, ε, της συνεργασίας ε, μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων σε επίπεδο Βρυξελών, από την έδρα των Βρυξελών. Ε, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει εγώ να συνεχίσω τις προσπάθειες για να μπορέσω ε, να προωθήσω τα θέματα για την διαχείριση κρίσεων και άλλα. Στην πρώτη μας συνεδρίαση είχαμε μία κοινή συνεδρίαση με τους υπευθύνους ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να συζητήσουμε συζητήσουμε ορισμένα θύματα. Σας είπα ότι ε, στις 16 ε, Φεβρουαρίου θα συζητήσουμε και με τους γεωγραφικά προσκύμενους συναδέλφους για τα θέματα της, Μέσων, της Μέσης Ανατολής και ε, για να υπάρχει και στενότερη συνεργασία μεταξύ ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου μας. Επίσης προσπαθούμε να συντονίσουμε τις εργασίες ε, ε, και τις διαβουλεύσεις κατά τρόπον ώστε να προχωρούμε πιο επικοδομητικά. Βέβαια αυτό που είναι βασικό είναι η εσωτερική και εξωτερική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αυτό συζητήθηκε και στα προηγούμενα θέματα της Μερσίας Διατάξεως κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την ενίσχυση της αρχιτεκτονικής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την ε, συνθήκη της Λισαβόνας για να συνεργαστούμε καλύτερα με τους ε, διάφορους οργανισμούς που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και μας ενδιαφέρει να ενημερωθούμε για τα μαθήματα τα οποία μπορούμε να αποκομίσουμε από τις σχέσεις μεταξύ αυτής της Επιτροπής και της Επιτροπής Ελευθεριών παραδείγματος χάρη που παρακολουθεί παρεμφερή θέματα. Ουσιαστικά όμως έχουμε ε, δύο θέματα αφενός η ε, εξωτερική υπηρεσία πρέπει να εντύπωσε Τη της να μπορέσει να αναλάβει τις ευθύνες της ε, ε, ε, να συντονίσει με τους γεωγραφικούς εκπροσώπους που συμβάλλουν σε αυτές τις συζητήσεις. Επίσης, ε, παλιά είναι και θέμα προσωπικού. Προηγουμένως συζητούσαμε ε, με τρεις ομολόγους από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ενώ τώρα έχουμε μόνο έναν που είναι η υπηρεσία εξωτερικής εξωτερικής δράσης. Ε, όσον αφορά την ε, οριζόντια και κάθε τη κατανομή ε, των δράσεων για το διάλογο θα πρέπει όλα αυτά να τα εξετάσουμε πολιτικά. Από πλευράς πολυμερού είπαμε ήδη για την αναθεώρηση του Συμβουλίου που θα είναι ένα πολύ βασικό θέμα που θα μας απασχολήσει ε, η προετοιμασία και της Γενικής Συνέλευσης για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας και να συντονίσουμε τις εργασίες μεταξύ Γενέβης και Νέας Υόρκης και ε, να είμαστε ε, έτοιμοι για τη συνεδρίαση της 16ης του μηνός. Επίσης, αν υπάρχουν θέματα για το επικείμενο συμβούλιο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε σε σχέση με ερωτήσεις. Γι' αυτό και εγώ τώρα δεν θα προσπαθήσω να αναφερθώ στις ε, προκλήσεις που δημιουργεί κάθε προτεραιότητα και κάθε καθευθυντήρια γραμμή διότι θα ε, προτιμώ να κερδίσω περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση που θα έχουμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρεσβευτά. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στα μέλη της υποεπιτροπής. Ποιος θέλει το λόγο? Η κυρία Μπάρμπαρα Λόχμπιλερ. Thank you, uh, Mr. Chair. I think... Ευχαριστώ. Δεν ε, έχουμε και πολλά να σχολιάσουμε διότι ήταν ε, εξαντλητικός ο κατάλογος των όσων μας ανέφερε. Θα μπορούσε λοιπόν να μας ε, δώσει τη σημειώση του γιατί δεν προλάβαινα να τα καταγράψω όλα. Αυτό που έχει σημασία είναι να ασχοληθούν με τα ατζέντα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε κάθε σύνοδο βλέπουμε ότι δεν ε, πετυχαίνουμε τους στόχους μας Είπατε ότι θα εντατικοποιήσετε τις προσπάθειές σας ε, και θα θέλαμε να ακούσουμε από εσά ε, και πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά και για τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος μας, η κυρία Χάουταλα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Οι ψυχολόγοι μιλάνε για γνωστική έλλειψη συντονισμού και νομίζω ότι ακούγοντας ε, τον πρέσβη διάβαζε το πρόγραμμά μας. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει μια πιο στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στον ε, ΚΟΧΟΜ και την Επιτροπή μας. Πώς όμως ε, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την ε, λιγότερη διαφάνεια η οποία ενδέχεται να προκύψει μετά από τις ε, από την ε, σύσταση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κάποια ζητήματα κλειδιά και θα ήθελα να δούμε πώς θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε και να βοηθήσουμε τόσο το Συμβούλιο όσο και την ύπαντη ε, εκπρόσωπο. Εμείς ως υποεπιτροπή χρειάζεται να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες και φυσικά κατανοώ απόλυτα την ανάγκη των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες αλλά ορισμένα έγγραφα είναι τέτοιας φύσης που δεν μπορούν να δημοσιοποιούνται ως εκ τούτου χρειάζεται να βρούμε ένα είδος συνύπαρξης ή κοινή κατανόησης το πώς η Επιτροπή μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάποιες στρατηγικές φύσεις πληροφορίες. Παράδειγμα, σήμερα έγραψε μια επιστολή, α, σε ποιον, α, ναι, ναι, στην κυρία Άστον. Ξέρετε, γράφω τόσο πολλές επιστολές που μπλέκομαι μια φορά. Και τη υπενθυμίζω ότι η κυρία Λόχμπιλερ έκανε μια ερώτηση για τον αποκλεισμό πώληση όπλων στην Κίνα. Θα ενθυμίστε την συζήτηση που είχαμε όπου μας είπατε ότι η συζήτηση ήταν το θέμα μάλλον ιδιαίτερα πολιτικού χαρακτήρα και ήταν δύσκολο για σας να απαντήσετε. Θα θέλατε να σας κάνουμε πιο, πιο απτές ερωτήσεις factual και σας ρώτησα τι εννοείτε. Ξέρω ότι υπάρχουν δύο φάκελοι που ένας αφορά την Κίνα, ο άλλος την Ρωσία και τις σχετικές πωλήσει όπλων. ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε μια φιλική διευθέτηση του ζητήματος ε, με την κυρία Άστον και τα μέλη του Συμβουλίου για το θέμα αυτό των πληροφοριών. Και κάτι ακόμα που θίξατε μεταξύ των πολλών δηλώσεων που κάνετε είναι αυτή η διαφορά ανάμεσα στις εσωτερικές, τις πολιτικές, τις εσωτερικές και τις εξωτερικές. Έγινε αναφορά στο θέμα των ε, παραδόσεων ε, της CIA. Ξέρετε το θέμα είναι λεπτό, δεν είναι διόλου εύκολο να εξεταστεί ακόμα και στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Υποεπιτροπή ελπίζουμε ότι θα έχει μια στενή συνεργασία με την ε, επί της Αρμόδια Επιτροπή, την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Χρειάζεται λοιπόν να συνεχίσουμε εμεί στην υποεπιτροπή μας να εξετάζουμε το θέμα αυτό, διότι πολλά τρίτα κράτη έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει το πρόβλημα της ατιμορρησίας. Και θα ήθελα να σας θέσω κύριε Τόγεμαν αυτή την ε, πολιτική φύση ερώτηση. Βλέπετε πως ε, στο εγγύς μέλλον ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, θα ασχοληθεί με το ζήτημα. Ξέρουμε ότι έχουν διαρρεύσει πολλά μέσω του Wikileaks, κάτι το οποίο βεβαιώνει ε, αυτό που είχε συμπεριλάβει το Κοινοβούλιο στην ε, έκθεση του 2007. Δεν αφορά μόνο ζητήματα κυριαρχίας κατών μελών, αλλά είναι κάτι που αφορά άμεσα την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε να κηρύττουμε την ε, ατιμορρησία. Θα έρθει λοιπόν κάποια μέρα όπου τα ζητήματα αυτά θα εξεταστούν. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Θέλει άλλος κανείς το λόγο. Ε, ε. Κι εγώ κύριε Πρέσβη θα ήθελα να σας ε, θέσω μια ερώτηση, γιατί πραγματικά είστε σε ένα οριακό τομέα, γιατί έχουμε πολύ έντονα οικονομικά συμφέροντα από τη μία πλευρά, αλλά και το πολύ σημαντικό γεγονός ότι όλος ο κόσμος προσπαθεί να ανακάμψει από την κρίση, ε, υπάρχουν τα εμπορικά ζητήματα, υπάρχει συνεργασία με τους στρατηγικούς μας τέρος και όλα αυτά τα θέματα προβάλλονται ιδιαίτερα. Βέβαια έχουμε και τεράστια συμβολή σε αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Αναφέρθηκαν και κατοχυρώθηκαν τα νέα αυτά όργανα και μηχανισμοί. Πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα μέσα αποτελεσματικά ώστε να έχουν θετικά αποτελέσματα και να μας, αποφέρουν, να μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε τους στόχο μας. Η πολιτική συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προαγωγή των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων καλό θα ήταν να συνδυαστεί και με τι υπόλοιπε πολιτικέ. ώστε να μην έχουμε μια αμυγή διαδικασία προώθηση και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία, αλλά μια πολιτική που θα συνδυάζεται με την ανθρωπιστική βοήθεια, με την οικονομική πολιτική, με την εμπορική πολιτική. Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε εύκολα να χρησιμοποιήσετε τα θετικά αποτελέσματα συνεργασίας με τους υπόλοιπους εταίρους με τους οποίους θα έχετε όλες αυτές τις συζητήσεις και θα μπορούσατε εκεί να συνδέσετε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις άλλες πολιτικές. Δεν βλέπω άλλο βουλευτή να ζητά το λόγο, γι' αυτό θα σας ε, δώσω το λόγο για την απάντηση, κυρία Πρέσβευτα. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και για τις ερωτήσεις σας. Επαναλαμβάνω ότι για μας η δική σας υποεπιτροπή είναι ένας πολύ φυσιολογικός, ε, φυσικός εταίρος μας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους ε, υπερμάχους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλά συμβάλλει σε αυτό το θέμα η Επιτροπή σας αλλά και το Συμβούλιο. Γι' αυτό και θα έχουμε στενή συνεργασία και προβλέπουμε σε μια τέτοια στενή συνεργασία, ώστε πραγματικά να συσπυρώσουμε τι προσπάθειές μα για να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Όχι μόνο για του ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και για όλα τα θέματα στα οποία θα συνεργαστούμε. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και την πρόσβαση στι πληροφορίε, το ζήτημα αυτό όντω είναι σημαντικό. Το είπατε κι εσεί ότι ορισμένα από τα έγγραφα και κάποιε στρατηγικέ που επεξεργαζόμαστε για τις στρατηγικές, για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάποιες έρευνες που γίνονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πάντα προβληματιζόμαστε θα πρέπει να δημοσιεύονται και πολύ συχνά ε, επιλέγουμε την εμπιστευτικότητα. Γιατί αν είναι να δημοσιευθούν αυτά τα έγγραφα, θα είναι πολύ πιο διπλωματική η διατύπωσή τους. Πάντως σίγουρα χρειάζεται εντατική συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας και για το θέμα της πρόσβασης στα έγγραφα. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό, όχι μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί προσπαθεί αυτή τη στιγμή να εναρμονίσει τους κανόνες για τη διαφάνεια, την πρόσβαση στα έγγραφα και πριν από λίγες μέρες έγινε μια συνάντηση μεταξύ της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και του Κοινοβουλίου για την ε, πρόθεση αυτής της διαδικασίας και θα υπάρξει εξέλιξη σύντομα. Πάντως και στο παρελθόν προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε για το θέμα αυτό, αλλά ότι σε ό,τι αφορά την ανάλυση των πληροφοριών, ε, εν ώψη συναντήσεων, διαλόγων διαβουλεύσεων θα συνεχίσουμε τη μέχρι τώρα πολιτική μας, να ενημερώνουμε τη γραμματεία σας για αυτές τις προσπάθειες, να σας δίνουμε τα χρονοδιαγράμματα ή να σας ενημερώνουμε και κλεισμένο το θηρό για τις διαβουλεύσεις που κάνουμε. Και θέλουμε να βελτιώσουμε και να καταστήσουμε πιο αποτελεσματικές αυτές τις ανταλλαγές. Πολλές ερωτήσεις τέθηκαν για το θέμα συνάφειας μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Εγώ ε, προηγουμένως είχα ασχοληθεί με την εσωτερική διάσταση και μάλιστα προσπάθησα την ε, ad hoc ομάδα εργασία για τα θεμελιώδη δικαιώματα να τη μετατρέψω σε μια μόνιμη ομάδα εργασία με ισχυρή εντολή. Γιατί αυτό το θέμα για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και προσφυλέ. Και στο Συμβούλιο σημειώθηκε πρόοδο, αλλά μόνο το τελευταίο εξάμεινο έγιναν σοβαρέ συζητήσει ότι για πρώτη, και για πρώτη φορά η Κοχόμ είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της, ε, του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, κάτι που στο παρελθόν δεν είχε γίνει. Και στο φόρουμ των μη κυβερνητικών οργανώσεων έγινε για πρώτη φορά λόγος για το θέμα αυτό. Σε όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της, εξωτερικής, ε, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, ό,τι αφορά τα πορίσματα προηγουμένων ε, εκθέσεων. για τις παράνομες απαγωγές της CIA. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το θέμα δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αλλά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε καλύτερα να επιληφθεί όχι η ΚΟΧΟΜ, αλλά η ομάδα εργασία για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και η ομάδα εργασία για τα θεμελιώδη δικαιώματα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη, στα Σπάργανα. Έχει νέα εντολή για το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά δεν έχει αναπτύξει ακόμη τη μεθοδολογία για να υλοποιήσει αυτή την εντολή. Επικεντρώνεται προ το παρόν η ομάδα αυτή εργασία στο θέμα τη προσχώρηση στην ε, ε, σύμφαση του, στη συνθήκη του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα θα έχουμε και την ετήσια έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θα αναπτυχθεί σταδιακά αυτή η νοοτροπία, αυτή η κουλτούρα ε, για την ε, συζήτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διάφορες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως εμείς, η ΚΟΧΟΜ, έχουμε μια εντολή που είναι αμυγός εξωτερική και θέλουμε στενή συνεργασία με την ομάδα εργασία θεμελιώδων δικαιωμάτων, γιατί θα υποφεληθούμε και εμεί από αυτή. Σε διαβουλεύσει και διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και σε πολυμερή φόρα, πολύ συχνά προσκρούμε σε συζητήσει για την κατάσταση εντό Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να μπορούμε να έχουμε και εμεί λόγο για τα θέματα αυτά. Έγιναν κάποιες ερωτήσεις για το πώς θα καταστήσουν πιο αποτελεσματικά τα αναπτυξιακά μας μέσα σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Μέσο Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτή τη στιγμή διενεργούνται διάφορες μελέτες επιπτώσεων για να δούμε πώς λειτουργούν αυτά τα μέσα. Αλλά ίσως για αυτό το θέμα θα ήθελα να προσθέσει κάτι ο συνάδελφος ή η συνάδελφοι. Επίσης, συνεργασία ή μάλλον διαπλοκή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με άλλες ε, πολιτικές. Όπως ε, προβλέπεται στη συνθήκη της Λισαβόνας, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα είναι πια ένα μεμονωμένο ζήτημα, αλλά θα πρέπει να είναι ένα απόσπαστο τμήμα τη συνολική πολιτική μα απέναντι σε τρίτε χώρε. Και αυτό το θέμα τη ε, ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκέ πολιτικέ θα βρεθεί στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων. Καλό θα είναι σε πρώμο στάδιο και με συνεπή τρόπο να καταστήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα αναπόσπαστο τμήμα των ευρωπαϊκών πολιτικών για να επιτύχουμε αυτή τη συνέπεια και τη συνοχή που επιδιώκουμε και αυτό φυσικά θα το αναλάβει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ως ε, θεσμό, ως θεσμικό όργανο, ε, γιατί έχουμε και εμείς σχετική εμπειρογνωμοσύνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα εξασφαλίσουμε συμπερίληψη τους σε ευρωπαϊκές πολιτικές, αλλά και η ΚΟΧΟΜ μέσω των γεωγραφικών της ε, γραφείων και μέσω της συνεργασίας με τις ομάδες εργασίας που βρίσκονται σε διάφορες ζώνες του κόσμου θα εξασφαλίσουμε αυτή την ε, προσπάθεια για την βελτίωση του συστήματος, γιατί η COHOM δεν θα πρέπει να είναι μια απομονωμένη ομάδα εργασίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, αλλά είναι ένα απόσπαστο τμήμα αυτής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση που μας κάνατε και φυσικά πολύ ενδιαφέρουσες και απαντήσεις ε, που μας δώσατε. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος να λάβει το λόγο για το σημείο αυτό. Όχι. Οπότε θα προβούμε σε δεκάλεπτη διακοπή πριν περάσουμε στην κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Αντιπροσωπεία για το Μαγκρέπ για την Τινησία. Σας ευχαριστώ. Ε, Συγγνώμη, μια σημαντική ανακοίνωση πριν φύγετε. Ο Αντιπρόεδρος Ξύπ και εγώ αύριο θα οργανώσουμε μία συνεδρίαση που οργανώνει το Λαϊκό Κόμμα με θέμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την ελευθερία έκφραση στο Καζακστάν. Θα γίνει μεταξύ 3 και 4 στο 3, στην αίθουσα σε. Υπάρχει τελευταία έντονα ενδιαφέρον για το Καζακστάν, γι' αυτό παρακαλείστε όλοι αύριο στις 3 με 4 στην ακρόαση που θα διοργανώσει το ΕΛΚ για το Καζακστάν.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 Καλωσορίζοντα σας ε, στην κοινή συνεδρίαση. Από τις 6.30 και μετά θα έχουμε μόνο αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά και πολωνικά. Μέχρι τις 6.30 έχουμε όλες τις γλώσσες, αλλά από τις 6.30 και μετά θα έχουμε λιγότερες γλώσσες. Περνάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης, που Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ξεκίνησε σήμερα στις 3, αλλά αυτό το κομμάτι γίνεται από κοινού με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Αντιπροσωπεία για τη σχέση με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέπ. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα στην κοινή μας συνεδρίαση και ελπίζω λίγο αργότερα να έρθει και ο κύριος Αλαφράγκα, ένας από τους δύο συμπροέδρους της Αντιπροσωπείας και μέχρι τότε έχουμε μαζί μας τον κύριο Παντσέρη, τον δεύτερο αντιπρόεδρο της ε, αντιπροσωπείας για το Μαγκρέπ και βλέπω και πολλά μέλη της ad hoc αντιπροσωπείας, τον κύριο Μπουσουτήλ για παράδειγμα, την κυρία Ρομέρο Λόπες, την κυρία Σενκλέρ. φάνηκε ότι ήταν και κάποιον άλλον από την ad hoc αντιπροσωπεία. Α, και εγώ που εκπροσωπώ την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Αντχόκ Αντιπροσωπεία. Η Αντχόκ Αντιπροσωπεία επέστρεψε λίγο πριν από την Τινησία. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με σχεδόν όλους τους ε, βασικούς φορείς ε, αυτής της μετάβασης που λαμβάνει η χώρα στην Τινησία και νομίζω ότι όλοι εστερνιζόμαστε την ειλικρινή επιθυμία και ελπίδα ότι οι πολίτες της Τινησίας θα απολαύσουν ένα γνήσια δημοκρατικό σύστημα με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, απόλυτη επικράτηση του κράτους δικαίου. Εγώ έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε μια μοναδική πραγματικά κατάσταση. Δεν νομίζω ότι είχαμε παρόμοια εμπειρία. Είναι άνευ προηγουμένου αυτή η πρόκληση. Γιατί βέβαια η, νησία, η Τινησία σε καμία περίπτωση δεν ήταν κράτος αποτυχημένο, άναρχο, άνομο και έχει όλα τα θεσμικά όργανα, έχει όλα τα θεσμικά όργανα που χρειάζεται ένα δημοκρατικό κράτος. Απλώς ε, ε, όλα αυτά τα θεσμικά όργανα για 23 χρόνια ήταν έρμεα ή ήταν όμοιροι μάλλον μιας ε, αδίστακτης δικτατορίας που χαρακτηρίστηκε από μεγάλη κατάχρηση εξουσίας από τον πρόεδρο και μια, ένα μικρό αριθμό οικογενειών που ασκούσαν την εξουσία ουσιαστικά. Και μάλιστα σε διεθνείς οργανώσεις υπάρχει μεγάλη προθυμία για να τίνουμε μια χείρα βοηθεία προς την Τινησία προκειμένου να διέλθει αυτή τη δύσκολη μεταβατική περίοδο. Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, από τους πιο σημαντικούς φορείς της υποστήριξης αυτής και υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες προς εμάς. Πολλές φορές ακούσαμε από ομολόγους μας ε, από την Τινησία ότι η χώρα αυτή έχει πλούσιο δυναμικό, δεν θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί εκ βάθρων. Αυτό που χρειάζεται είναι συγκεκριμένη ουσιαστικά βοήθεια, μια συμβουλή, συγκεκριμένες τεχνικές συμβουλές και ελπίζω η υποστήριξη αυτή η βοήθεια ε, προς την Τινησία να δρομολογηθεί με σωστό τρόπο από την διεθνή κοινότητα για να μπορέσει η χώρα αυτή να αξιοποιήσει αυτή την διεθνή υποστήριξη. Οπότε ξέρω αύριο στην Τίνιδα θα συναντηθούν Ευρωπαίοι πρέσβεις με την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία για να συζητήσουν όλα αυτά τα θέματα και εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στενά με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΟΗΕ και με την Επιτροπή της Βενετίας που είναι αξιοθαύμαστος σύμβουλος για θέματα συνταγματικά και γενικώ υπάρχει όλη αυτή η τεχνογνωσία που χρειάζεται σε αυτούς τους μεταβατικούς καιρούς. Αυτά προς το παρόν από μένα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Παντζέρη, που είναι ο συμπρόεδρος της Ατχόκ Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Τινησία, για να μας παρουσιάσει τις ε, εμπειρίες που είχαμε εκεί και τις απόψεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν συντομία, θα σας αναφέρω τι κάναμε και ορισμένες εντυπώσεις μου. Εξάλλου έχει διανυμηθεί το ανακοινωθέν τύπου το οποίο εκδώσαμε που είναι αρκετά εύγλωτο σχετικά με τα αποτελέσματα που διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, επίσκεψη την οποία πραγματοποιήσαμε όταν ακόμα η κατάσταση ήταν πολύ περιπεπλεγμένη ήρεμη μεν, αλλά περιπεπλεγμένη, δε από πολιτική σκοπιά αλλά και από πλευρά ασφάλεια. Κατά τη διάρκεια τη παρουσία μα στην Τινησία έγιναν πολλέ διαμαρτυρίε και δυστυχώ τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή του και όσα αντιπροσωπεία καταγγείλαμε τα όσα συνέβησαν. Το πρόγραμμά μας ήταν ιδιαίτερα πυκνό και μα επέτρεψε να γνωρίσουμε εκ του σύνεγγυς την κατάσταση μετά από την απομάκρυνση του πρόεδρου Μπέναλή και ήταν επικοδομητική επίσκεψή μας ξεκινώντας από τη συνάντηση που είχαμε με τι τρει επιτροπέ οι οποίε συγκροτήθηκαν μετά από την ε, πτώση του Μπέναλή ε, Επιτροπή για την Πολιτική Μεταρρύθμιση την Επιτροπή κατά της διαφάνειας και των επεξαιρέσεων και η Επιτροπή η οποία θα έπρεπε να εξετάσει τις εξελίξεις και τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν. Οι λοιπόν που είχαμε αυτές τις επιτροπές, ειδικά με την Πολιτική Επιτροπή και τον πρόεδρο της Μπένα ε, ένα πρόσωπο το οποίο είναι ιδιαίτερα γνωστό και αναγνωρισμένο από τους Τινήσιους. Ε, μας ε, ξέθεσε λοιπόν πως η κατάσταση είναι ρευστή. Ο κύριος ο ίδιος ο πρόεδρος Μπένα Σούρ μας είπε ότι ξεκινάει μια φάση διαβούλευσης με τις πολιτικές δυνάμεις, με την κοινωνία των πολιτών, με, τις, ε, με όλες τις κοινωνικές ομάδες ε, και για να δουν τι στρατηγική πρέπει να εφαρμόσουν για να βγουν από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η χώρα αυτή. Βρισκόμαστε ε, παρουσία μιας προσωρινής κυβερνήσεως η οποία δεν είναι ακόμα αναγνωρισμένη είναι ιδιαίτερα αδύναμη θα έλεγα αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ως συμπέρασμα της συνάντησής μας είναι η εντύπωση ότι αυτός ο Πρωθυπουργός ήταν μόνος του σε αυτό το προεδρικό κτίριο η κατάσταση λοιπόν είναι πολύ λεπτή και θα πρέπει να, να διαπιστώσει συγγνώμη, ποια θα είναι η στρατηγική που χρειάζεται να προωθήσει την Ισία για να ολοκληρώσει τις ε, θεσμικές αλλαγές ε, κλπ. Αυτή είναι η εντύπωση που είχαμε όταν συζητήσαμε την Πολιτική Επιτροπή αλλά και άλλους από πού θα πρώτο ξεκινήσουν διότι η ιδέα που επικρατεί από πλευράς τουλάχιστον Προέδρου της Πολιτικής Επιτροπής είναι να φτάσει στις προεδρικές εκλογές με βάση το ισχύον σύνταγμα. Κάτι που από ορισμένες πλευρές παρουσιάζει μια κάποια νομιμότητα αλλά συνάμα και κάποια προβλήματα διότι το ισχύον σύνταγμα είναι ένα σύνταγμα ανελεύθερο και κινδυνεύουμε να έχουμε εκλογή Προέδρου της Τινησίας ε, νομοποιημένου από το λαό αλλά που θα στηρίζεται σε, μια, σε ένα σύνταγμα το οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί, να μεταρρυθμιστεί και δεν ε, σημαίνει ότι ο Πρόεδρος θα κάνει αυτή την μεταρρύθμιση της αλλαγές με τον ε, πιο σωστό και κατάλληλο τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια συντακτική βουλή και μετά να ξεκινήσουν ε, εκλογές να δουν κατά πόσον ο τυνησιακός λαός θέλει να έχει μια προεδρική δημοκρατία ή μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτό είναι ένα κομμάτι της συζήτησης που δεν έχει γίνει προς το παρόν. Υπάρχει λοιπόν μια τάση, μια έθεση να συσταθούν ε, τα κόμματα, να μπορέσει να ξεβρεθεί μια κάποια ημερομηνία. Από ό,τι κατάλαβα, δεν ξέρω αν και τα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας ε, κατάλαβαν το ίδιο, δηλαδή μιλάμε για μια περίοδο ενός εξαμήνου προκειμένου να φτάσουν στις ε, προεδρικές εκλογές στην Τινησία. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι μια συζήτηση που ακόμα είναι ανοιχτή, εκκρεμή. Θα επανέλθω αργότερα για να εκφράσω την προσωπική μου άποψη, αλλά προς το παρόν αυτά κατά έχουμε καταλάβει. Συναντήσαμε κάποια μέλη της προσωρινής κυβέρνησης ε, και αυτές οι συναντήσεις είχαν ιδιαίτερη σημασία διότι μας επέτρεψαν να κατανοήσουμε ποια είναι η τάση που θέλει να ακολουθήσει ε, αυτή η κυβέρνηση. με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με τον οποίο εξετάσαμε το ζήτημα έρθμιση της δικαιοσύνης και της ανεξαρτησίας ε, του δικαστικού κλάδου. Είχαμε μια συνάντηση πολύ ενδιαφέρουσα με τον Υπουργό Άμυνας. Όπως γνωρίζετε, το στράτευμα είναι ο μοναδικός ε, θεσμός ε, τον οποίο αναγνωρίζουν οι πάντες στην ε, την Ισία διότι είναι ένα όργανο που δεν επενέβη και εγγυήθηκε αυτή την μεταβατική περίοδο, τη διαδικασία μετάβασης. Είχαμε μια σημαντική συνεδρίαση συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών ο οποίος μετά από μια αναλυτική συζήτηση για το μέλλον της Τινησίας μας ε, ενεχειρίασε και μια επιστολή προς το Ευρωκοινοβούλιο προκειμένου να δώσουμε την συμβολή μας για αυτές τις διαδικασίες. Επίσης συναντήσαμε και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας των πολιτών. Αναφέρομαι στην οργάνωση των δικαστικών, τον ε, δικαστικό, δικηγορικό σύλλογο, συγγνώμη, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν συνάντηση με το Ισλαμικό κόμμα. Κάνα μια σειρά παρατηρήσεων και σχόλια, δηλαδή το πώς βλέπουν το μέλλον της Τινησίας και πραγματικά μας απάντησαν αναλυτικά με βάση δημοκρατικές αρχές και να πω εδώ ότι το Ισλαμικό κόμμα μας ε, ε, έβαλε ένα αίτημα εάν ε, απέναντι σε μια στην περίπτωση που το Ισλαμικό κόμμα ε, πάρει την πλειοψηφία στις ε, εκλογές τι θα κάνει η Ευρώπη γνωρίζοντας ποια είναι τα αποτελέσματα με τις εκλογές που έγιναν στην Παλαιστίνη και τις εξελίξεις εκεί. Εμπεστώς είχαμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση που μας επέτρεψε να καταλάβουμε ότι Υπάρχει μια <clears throat> κάποια αναταραχή, υπάρχουν ορισμένα κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή συγκροτούνται δεν έχουν ε, λάβει ακόμα την άδεια προκειμένου να ε, συγκροτήσουν το κόμμα. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα πτυχή διότι στην αξιολόγηση που μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με την ισιακή ε, πραγματικότητα είναι ότι η κοινωνία των πολιτών κατά κάποιο τρόπο ξεπέρασε όλα τα θέματα που αφορούσαν ε, την, <clears throat> την περίοδο Μπέναλη, αλλά θα πρέπει τώρα να συσταθούν, να συγκροτηθούν τα πολιτικά κόμματα, διότι αποτελούν τη ρεχοκοκαλιά μιας δημοκρατικής διαδικασίας ε, στην Τινησία και με την κοινωνία των πολιτών. Λοιπόν, η συζήτηση ήταν πολύ σοβαρή και μας επέτρεψε να κατανοήσουμε τα άγχη, τις προσδοκίες. Διεξάγεται συζήτηση και μεταξύ τους, αλλά όχι μόνο μεταξύ τους, κατά πόσον θα πρέπει να προχωρήσουμε με την εκλογή του Προέδρου ή αν θα πρέπει να συσταθεί ένα επαναστατικό συμβούλιο το οποίο θα παρακολουθεί τα τεκτενόμενα μετά από τις ε, εξελίξεις, μετά από την επανάσταση θα λέγαμε. Και στην Τινησία υπάρχει ένα θέμα το οποίο <clears throat> κυριαρχεί και αυτό προέκυψε στις συζητήσεις ε, και με την κοινωνία των πολιτών και με το δικαστικό σώμα και με τον δικηγορικό σύλλογο αλλά και με τους δικηγόρους. Μια ε, σοβαρή κριτική, μια στεναρή κριτική απέναντι στην Ευρώπη, την οποία πρέπει, στην οποία εμείς πρέπει να τίνουμε δίκον ούσου και η οποία έχει ως εξής, λέγοντας ότι εσείς κατά κάποιο τρόπο βοηθήσατε το καθεστώς του Μπέναλη και θα πρέπει να λογοδοτήσετε για ποιο λόγο δεν ε, κατανοήσατε εγκαίρως ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά στην και γιατί θα έπρεπε να υπάρξουν εξελίξεις. Σα είπα λοιπόν, οι συναντήσει ήταν πολύ σημαντικέ, πολύ επικοδομητικέ, αλλά και πολύ σκληρέ σε κάποιες περιπτώσεις. Κατα, καταλήγω λέγοντα ε, ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να συναγάγουμε από αυτή την επίσκεψη. Το συνέστημα, το οποίο πιστεύω ότι συμμεριζόμαστε όλοι, και ελπίζω τουλάχιστον, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κάπως συγκεχημένη. Υπάρχει ένα ε, αντικειμενικό στοιχείο που είναι η προετοιμασία και ο τρόπος προετοιμασίας, αλλά πέραν των τριών των επιτροπών που προανέφερα, ε, δεν υπάρχει κάποιος χώρος όπου ε, τα διάφορα εμπλεκόμενοι μπορούν να συναντήσουν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σχετικά με την ε, ιδέα μιας επιτροπής η οποία θα μπορέσει να προχωρήσει σε συνταγματικές αλλαγές, θεσμικές αλλαγές κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να οικοδομηθούν. Άρα υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει ένα κενό εξουσίας. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες ε, συγκρούσεις, ε, υπάρχουν κάποιες ε, καταγγελίες, υπάρχει ακόμα το μεγάλη κλίκα των εισαγωγικών του Μπέναλή που δράσε όλη την επικράτεια και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Τώρα τα θεμελιώδη προβλήματα τα, τα απαριθμώ, δεν τα ερμηνεύω. Οικονομική και δημοσιονομική κρίση. Κρίση στον τομέα του τουρισμού. Και ενδεχόμενα αυτό να οδηγήσει σε μια περαιτέρω χρέωση από πλευράς ε, την Ισίας. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της ασφάλειας, ασφάλειας των προσώπων, των ε, θεσμών, αλλά και του οικονομικού και παραγωγικού συστήματος, παραγωγικού ιστού. Και ένα ακόμα τρίτο πρόβλημα είναι δημιουργία της δημοκρατικής διαδικασίας, τι μεταρρυθμίσεις, ε, μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης, ε, ε, η ελευθεροτυπία και το ζήτημα των ελευθεριών εν γέννη. Μιλάμε για αστικές ελευθερίες, άρνηση, θρησκεία κλπ. Και Ολοκληρώνω λέγοντας ότι για να βοηθήσουμε αυτή την ε, μεταβατική περίοδο, μεταβατική διαδικασία, να ε, εφαρμόσουμε το προωθημένο καθεστώς. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο οικονομική και κοινωνική συνεργασία και ένα στήριγμα στην κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει να συζητήσουμε το ζήτημα της μετανάστευσης και των ε, ε, στοχευμένων ε, παρεμβάσεων διότι αυτή είναι μια βαλβίδα ασφαλείας ε, που δεν υπάρχει ειδικά σε ό,τι αφορά την με, μετανάστευση ανθρώπων του πνεύματος και κάτι ακόμα το οποίο εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο προημερών υιοθετήσαμε το ζήτημα της Task Force για στήριξη στη δημοκρατική διαδικασία και τον εκδημοκρατισμό. Αυτό σημαίνει πως το Ευρωκοινοβούλιο μαζί με τα άλλα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Και ο τρόπος συμμετοχής προσωπικά πιστεύω ότι χρειάζεται να συμμετέχουμε όχι μόνο ως ε, παρατηρητές σε εκλογές, αλλά ευθύ αμέσω θα πρέπει να εγκατασταθεί μόνιμος. Να υπάρχει δηλαδή μόνιμη παρουσία. Εξάλλου αυτό έχει ζητηθεί από τα υποκατάρτιση κόμματα και από την κοινωνία των πολιτών. Αυτό νομίζω ότι εάν <clears throat> παρέλειψα κάτι έχουν με στην αίθουσα κάποιους συναδέλφους που συμμετείχαν στην αποστολή και μπορούν να συμπληρώσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε Παντσέρη για αυτήν την παρουσίαση και καλό τα μέλη της αντιπροσωπείας αν επιθυμούν να σχολιάσουν. Πάντως ε, θα ήθελα να τονίσω ότι ήδη στις Βρυξέλλες ε, ε, ο πρόεδρος Μπούζες συναντήθηκε με τον κύριο Γουένας και είχε δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται να αναχωρήσει από την νησία η αντιπροσωπεία χωρίς μία γραπτή πρόσκληση να παρακολουθήσουν σαν παρατηρητές εκλογές πράγμα το οποίο έγινε διότι θα πρέπει να είμαστε όχι σαν μία αποστολή παρακολούθησης αλλά θα έπρεπε να έχουμε και μακροπρόθεσμα κάποια παρακολούθηση για την εξέλιξη των συνθήκων στη χώρα αυτή διότι εγώ πρόσεξα ότι η κυρία Ρομέρο Λόπες ανέφερε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να οργανωθούν ελεύθερες εκλογές εάν υπάρχει μία τόσο ασαφής κατάσταση ασφαλείας ε, στην, ε, στην Ήπεθρο, σε, σε επίπεδο εκτός μεγάλων πόλεων. Οπότε πρέπει να δούμε πώς πρέπει να διατυπωθεί η πρακτική εμπλοκή του Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία και επειδή χρειαζόμαστε ενημέρωση γι' αυτό μας ενημέρωσε η εξωτερική υπηρεσία αλλά θα ήθελα να παρακολουσιάσω τον κύριο Τσεντουμπή πρόεδρο του Ευρωμεσογειακού Φόρουμ να μας ενημερώσει. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές. Εδώ σας ε, ομιλώ σαν ε, ελεύθερος άνθρωπος ο οποίος ξαναβρήκε την ελευθερία του και σαν πολίτης την Ίσιος αλλά και Ευρωπαίος διότι από την Ευρώπη και ιδιαιτέρως από τη Γαλλία όπου βρήκα φίλους πολυάριθμους οι οποίοι ε, συνέδραμαν τον τινησιακό λαό στον αγώνα του για την δημοκρατία. Ίσως δεν έχω επαρκή χρόνο για να εκφραστώ και γι' αυτό θα ήθελα να παρουσιάσω μία αναλυτική ε, ε, έκθεση ε, πήγα στην Τινησία μετά από 17 χρόνια ε, εξορίες και ελπίζω ότι θα μου δοθεί ο χρόνος να παρουσιάσω διάφορα στοιχεία τα οποία κατά την γνώμη μου είναι σημαντικά. Bien sûr, comme vous l'avez dit, la Tunisie entre dans une période de transition politique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 Thank you, Mr. Busuttil. You certainly reflect the sentiments we all had. So next I will give the floor to Mrs. Romero Lopez. Gracias, Presidenta. Quizá para dar alguna información complementaria, porque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 transition from dictatorship to democracy, because you certainly know how difficult and how challenging it is. But I give the floor to Vice Chair of the Subcommittee on Human Rights, Mr. Kazak. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est vrai que venant d'un pays qui aussi vient de passer une période de transition, il y a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 où tout va être décidé et on démocratique ait lieu et notre Parlement, notre Commission puisse avoir sa participation dans cette mission d'observation. Merci. Thank you very much for your remarks, Mr. Kazak. I have on my list Mrs. Ayala, who was also a member of the delegation, and Mr. Gahler. And I wonder if others present still want to take the floor, Mr. Mr. Zeller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 porque demuestra que los países árabes también se merecen la democracia y lo han sabido lo han sabido lograr por sí mismos. muchas gracias. Thank you, Mrs. Ayala. Now, I'm very pleased to invite Mr. Gahler to take the floor because he's the first who was not on this mission, but we very much expect him to say something in this debate